Good morning, dear colleagues. Good morning, everybody. Uh, ναι, να, ξεκινήσουμε την τακτική μας συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που προβλέπεται για σήμερα ως τις 12.30 και το απόγευμα από τις 3 έως τις 6.30. Και αύριο επίσης. Θα πρέπει να ανακοινώσω κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 7, ανακοινώσεις ε, της Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την δημιουργία επενδυτικού πλαισίου με τρίτες χώρες βάσει της Ευρωπαϊκής ε, Ατζέντα για τη Μετανάστευση 9 και 50 6 για την δικαστική συνδρομή για υπόπτωση κατηγορογμένου σε ποινικέ διαδικασίε και σε διαδικασίε εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Μετά το σημείο 8 στι 11.30. 13. Ερώτηση του Ιγνάτσιο Κοράου προ την Επιτροπή αναβάλλεται. 15 Κατάλογο των χωρών υπηκό των οποίων υπόκειται σε χώρε για και διέλευση των εξωτερικών και οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή κοσφοπέδιο σήμερα στις 12 αντί για αύριο το πρωί. Και προσθέθηκε ένα νέο σημείο στην εμείς διαταξή για αύριο το πρωί στις 9 για την κατάσταση κατεπήγοντος στη Γαλλία και την ε, συμμόρφωση αυτής με το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο τη Ένωση. Αυτά είναι τα, ε, οι χρονοθερίδες ενδεικτικά. Μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αντιρρήσεις προς την ημερήσια διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται για τις γλώσσες. Δεν έχουμε γελικά και κροατικά σήμερα και αύριο και η Ολλανδική διερμηνία δεν διατίθεται από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα. Πρέπει επίσης να δούμε θα εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών για, την, ε, για τον διορισμό συγητών, κυρίως τον κύριο Κύρκο, έκθεση για την ε, δημιουργία της Eurodac. Δεν θα διαβάσω όλα τα ονόματα. Η συγητής είναι ο κύριος Τίμωθη Κύρκο, προτείνεται δηλαδή. Ε, εγκρίνεται η σύσταση του συντονιστή μας. Θεωρώ πως ναι. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2015, 6 έως 9 Νοεμβρίου 2015, 17 Δεκεμβρίου 2015 και 20 έως 21 Απριλίου 2016. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στα πρακτικά, εγκρίνονται και αύριο, μάλλον τώρα, ξεκινάμε με τον κατάλογο τρίτων χωρών, η υπήκο των οποίων υποκεντρεί στην υποχρέωση θεωρήση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογο των τρίτων χωρών, η υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή να θεώρηση του μηχανισμού αναστολή. Η Επιτροπή πρότεινε το μηχανισμό αναστολή, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα κάποιες φορές να ζητάτε θεώρηση από τους κατοίκους των χωρών οι οποίες εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση. Ο κύριος Ντεμέρα είναι ο εισηγητής όταν είχε προβλεφθεί ο μηχανισμός αυτός αρχικά για τον κανονισμό. Να του δώσω ευθύ αμέσω τον λόγο. Κύριε Ντεμέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε για το μηχανισμό αναστολής. Όπως ε, σας είχα πει στις 26 Μαΐου, είναι μια έκθεση ε, προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για μένα. Οι διαπραγματεύσεις σημαντικών μέτρων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ουκρανία, το Κοσφοπέδιο, την Γεωργία και την Τουρκία εξαρτώνται από το αποτέλεσμα αυτού του, αυτού του εγχειρήματος. Οι πολιτικές επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις και οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις δεν πρέπει να λησμονηθούν. Ε, όπως παράδειγμα χάρη συμφωνία με την Τουρκία για το θέμα αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας τη στιγμή που θα προσπαθήσουμε να θέσουμε, να δρομολογήσουμε όλη αυτή την ε, προσπάθεια. Εγώ σας παρουσίασα ήδη το σχέδιο έκθεσης όταν με διορίσατε εισηγητή. Επίσης μίλησα με την Προεδρία του Συμβουλίου, μίλησα με την Κομισιόν και μίλησα με τους κοιόδης εισηγητές. Έχω υπόψη μου όλα τα στοιχεία και θα προσπαθήσω με αποφασιστικότητα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, αλλά και με ταπεινοφροσύνη, ούτως ώστε η έκθεση αυτή να είναι ικανοποιητική. Ο μηχανισμός αναστολής είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχει επιπτώσεις κυρίως στους υπηκόους τρίτων χωρών, με, τους οποίους η Ευρωπαϊκή, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες εξαίρεση από την υποχρέωση θεωρήσεων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες σε κάθε φάση της εφαρμογής ε, στην πρότασή μου ε, σας προτείνω να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό και γι' αυτό έχω βάλει τρεις βασικές ιδέες. Η πρώτη ε, συνδέεται με τις ε, κατεξιοδότηση Με βάση τον ισχύοντα μηχανισμό και την πρόταση της Κομισιόν, προβλέπεται ότι ο, η, λειτουργία αυτή ε, του όλου project θα γίνει μέσω ε, τέτοιων ε, πράξεων. Στην, στην πρότασή μου εγώ τις καταργώ και βάζω τις, ο, αποφάσεις με βάση τις οποίες θα εμπλακεί το Κοινοβούλιο, γιατί ούτως ή άλλως ως συνομοθέτης πρέπει να το κάνει. Αυτή είναι η θέση μου και την λέω με κάθε έμφαση. Θα πρέπει καταρχάς να τροποποιήσουμε ένα βασικό στοιχείο, μιας, ένας βασικού νομικού κειμένου. Αυτό γίνεται μόνο κατά εξουσιοδότηση πράξη και όχι μέσω εκτελεστικής πράξης. Η απόφαση του δικαστηρίου του 2015, της 16ης Ιουλίου του 2015, επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία. Ε, τη θεωρία με βάση την οποία εξέφρασε την απόψή μου. Όταν σας μίλησα για την, ε, το θέμα της αμοιβαιότητα, το οποίο αναφέρεται επίσης στην έκθεσή μου. Επίσης πρέπει να υπάρχει δια, ισοτιμία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το θέμα της ε, πολιτικής θεωρήσεων είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει να αποφασιστεί με την συνήθη νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Δεν έχει κανένα νόημα για να ε, αφαιρέσουμε την, τη θεώρηση από τρίτη χώρα και να την επαναφέρουμε, ή μάλλον ε, στην πρώτη περίπτωση συναποφασίζει και το Κοινοβούλιο, αλλά για να την επαναφέρουμε αποφασίζει μόνο το Συμβούλιο. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό δεν έχει κανένα νόημα για την κοινή λογική, αλλά και ούτε και νομική, νομική λογική έχει. Επίσης θα ήθελα να διασφαλίσουμε τις, ε, τα δικαιώματα των ε, υπηκόων τρίτων χωρών βάζοντας την ε, ανάγκη, μιλώντας για ανάγκη να είμαστε σοβαροί και αποτελεσματικοί. Ελπίζω αυτή η έκθεση να βελτιωθεί χάρη στις δικές σας ιδέες και κυρίως στις ιδέες ε, και τις ιδέες των σκιωδών εισηγητών, τις οποίες θα λάβω υπόψη μου στις τροπολογίες. Η προθεσμία για την παρουσίαση τροπολογιών θα είναι η 22 Ιουνίου και προτείνω να ψηφίσουμε στην Επιτροπή την επόμενη μέρα συγγνώμη, στις 12 Ιουλίου ε, προτείνω να ψηφίσει η Επιτροπή. Αυτά και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Διασταμέρα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τους κοιόδης ηγητές. Βλέπω την κυρία Γιώητοβα και θα της δώσω το λόγο. Και έχουμε βέβαια και τον εισηγητή της ΑΦΕΤ για το θέμα αυτό. και το κύριο Σάριους Βόλσκι, στον οποίο θα δώσω το λόγο, έχει έρθει για τη συζήτηση αυτή. Μπόνι, Σμίλα και Μπιόρκ στη συνέχεια. Ξεκινώ όμως με την κυρία Γιώτου. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πληρώσω κάποια λόγια στα όσα μας είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα. αφού τον ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ξέρουμε πως υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση παραβιάσεως από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Ορισμένοι από αυτούς τους μηχανισμούς δεν αξιοποιούνται. Επί έχουμε ακόμα αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το μηχανισμό αμοιβαιότητας της θεώρησης. Άρθρο 7 της συνθήκης. Και εδώ πάλι είναι αντιφατικό το κείμενο και θέλαμε από καιρό να επανεξεταστεί το άρθρο αυτό σε σχέση με την Πολωνία δεν συνέβη αυτό όμως. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητα δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ και αν ρωτήσει κανεί το γιατί, η Επιτροπή θα μας απαντήσει ότι δεν παρέστη ποτέ ανάγκη για κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως, τα μηνύματα που λαμβάνουμε δείχνουν πως μια τέτοια ενεργο, μια ενεργοποίηση τέτοιου μηχανισμού θα σήμαινε μεγάλο κόπο και διαδικασίες μακροσκελής. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο μηχανισμός και επιμένω. Πρώτον, θέλουμε να επιμείνουμε στην ε, χρήση των κατεξουσιοδότησης πράξεων και όχι των εκτελεστικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις σε αυτό το θέμα χωρίς ε, να λαμβάνεται υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι αυτή η αύξηση, η σημαντική αύξηση, είναι σκόπιμη. Μιλούμε για ένα ε, κατώτατο όριο του 50% για μια συγκεκριμένη περίοδο που όμως δεν είναι κατάλληλο διότι πολλά κράτη έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό υπηκών τρίτων ε, κρατών ε, τους τελευταίους μήνες. Επίσης θα πρέπει ο, οργανισ... ο μηχανισμός να ενεργοποιείται εάν δεν τηρούνται οι συμφωνίες. Και εδώ αναφέρομαι σε συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Εν τέλει, ο μηχανισμός κοινοποίησης είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει ε, κίνδυνος για την δημόσια τάξη. Πρέπει αυτό τον όρο να τον διευκρινίσουμε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα κλίμα καλή συνεργασία, αγαστή συνεργασία, και βέβαια πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση στο τέλο, Η πρόεδρο. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα. Μόλι έμαθα ότι η κυρία Μλίναρα την καθιστά τον κύριο Γέζεκ, οπότε να, σα σας, δώσω αμέσω το λόγο κυρία Μλίναρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Γέζεκ ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι καν εδώ. Οπότε σα μεταφέρω τι δικέ του θέσει και το μήνυμα του κύριο Γέζεκ στηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί ο μηχανισμός αναστολής θεωρήσεων βάσει των σημερινών εξελίξεων. Η κατάσταση τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόταση τη Επιτροπή για την Απελευθέρωση για την Ουκρανία και το Κωσυφοπαίδιο καθώ και την Τουρκία χρειάζεται να περάσει από ένα πιο εύρωστο και ρεαλιστικό πλαίσιο, ώστε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούν γρήγορα να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό σε περίπτωση που οι προποθέσει που θα ε, θέσουμε εμεί ε, θα καλύπτονται. Στην πράξη θα πρέπει να είναι και πιο προσαρμοσμένο το πλαίσιο αυτό στην πραγματικότητα και να είναι και πιο ευέλικτο. Επίσης καλωσορίζει τη συμπερίληψη της ανάγκης να δεχτούμε τις συμφωνίες επανεισδοχής. Όμως αυτή η αυξημένη ευελιξία πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες ε, εγγύησεις. Αυτές οι εγγύησεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα. Τελευταίο και εξίσου σοβαρό, δεδομένων των πολιτικών συνεπειών για την ε, νέα επιβολή των απαιτήσεων θεώρησης, ο κύριος Γεζίκ δέχεται την πρόταση του συγητή να συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο στη σχετική απόφαση και να ισχύει διαδικασία κατεξουσιοδότηση πράξεων, όπως προτείνεται στην έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Μλίναρ. Μόλις έμαθα ότι η κυρία Μπιόρκ αντικαθιστά την κυρία Βερζιά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μαρή Κριστίν μου ζήτησε να ε, τοποθετηθώ εγώ εκ μέρου τη. Οπότε έχω τι σημειώσει τις οποίες μπορώ να σας διαβάσω, αλλά θα μιλήσω γαλλικά για να προσπαθήσω να διαβάσω σωστά. Και να αλλάξουμε και λίγο η Μαρή Κριστίν υπογραμμίζει, αφού ευχαριστήσει τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε, γιατί εργάστηκαν μαζί, υπογραμμίζει για το μηχανισμό αυτό αναστολής στις σημερινές συζητήσεις και ιδίως ό,τι αφορά την Τουρκία, ότι θα πρέπει να προσέξουμε. Μην χρησιμοποιήσουμε τις πολιτικές θεώρησεις για να χαράξουμε πολιτικές και στόχους για τη μετανάστευση. Η πολιτική των θεωρήσεων δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο μέσο. Ένα δεύτερο σημείο που θέλει να θίξει είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Από τη μία και από την άλλη διαδικασία. Ως προς τα κριτήρια λοιπόν υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να είναι μόνο εργαλεία για να επιβάλλουμε μεταναστευτικέ πολιτικέ στα κριτήρια αυτά, οπότε είναι απαραίτητο το Κοινοβούλιο να απαιτήσει να υπάρχει απόδειξη τη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αγγίσεις για την πρόσβαση όλων στο δικαίωμα για άσυλο. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στα κριτήρια για την αναστολή και άλλα στοιχεία, όπω την κατάσταση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στι τρίτε χώρε, και δεν είναι λογικό ως κριτήριο αξιολόγηση για να δίνουμε το καθεστώ απελευθέρωση των θεωρήσεων τα δικαιώματα του ανθρώπου και όχι όταν κοιτάζουμε μήπω ανασταλεί ο μηχανισμό ή όχι. Ω προ το δεύτερο σημείο, τη διαδικασία, συμφωνούμε με τον εισηγητή Θέλουμε να γίνεται αυτό με κατεξουσιοδότηση πράξη, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Δεν είναι λογικό το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαδικασία για τι συμφωνίε απελευθέρωση και όχι όταν αναστέλλονται αυτές και τα σχετικά λόγματα. Αυτά. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν θυμάμαι πώς το λένε γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Ο, η κυρία Κίρκοπ, κύριος Κίρκοπ, θα μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Μακοβέη. Ε, θα σας δώσω το λόγο και μετά στον κύριο ε, Σάιρους Βόλσκι. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας εκφράσω τις απόψεις της κυρίας Μακοβέη. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες της. Αυτό που θέλει να ξεκαθαρίσει είναι ότι μιλάει για την ανάγκη ενίσχυση του μηχανισμού Αναστολή, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε μελλοντική και ισχύουσα ε, συμφωνία απελευθέρωση την υποχρέωση θεωρήσεων. Μια τέτοια ρήτρα αναστολή είναι σημαντική, ούτω ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε οποιαδήποτε κατεπίγουσα ανάγκη και επομένω να μην χρειαζόμαστε να περιμένουμε για μια λύση μέσω τη νομοθετική διαδικασία. Καλωσορίζει την πρόταση τη Κομισιόν, η οποία θα μειώσει την περίοδο αναφορά και τι προθεσμίε, ούτω ώστε η διαδικασία να είναι πολύ πιο γρήγορη και επεκτείνοντα του λόγου για του οποίου θα υπάρξει αναστολή. Ε, Δεδομένη τη σημερινή κατεπίγουσα κατάσταση, καλωσορίζει το, νέο λόγο για την ουσιαστική αύξηση των αριθμό ε, απορριφθισών αιτήσεων ε, από υπηκόους χωρών ε, που Είτε οι συμφωνίε επανεισδοχή έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από οποιοδήποτε κράτο ε, μέλο. Καλωσορίζει επίση την πρόταση του εισηγητή στην ε, τροπολογία 4 ε, που προσθέτει στον κατάλογο μία αύξηση ή πρόβλημα στην εθνική ασφάλεια ε, η δημόσια τάξη διαφωνεί με την τροπολογία 3 που επανεισάγει τη δυνατότητα ο μηχανισμός να χρησιμοποιείται μόνο σε κατεπίγουσες ε, περιπτώσεις, Πιστεύει και συμφωνεί με την πρόταση της Κομισιόν ότι ο μηχανισμός αναστολή θα πρέπει να χρησιμοποιείται πιο γενικά σε περίπτωση που η απελευθέρωση των θεωρήσεων οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της λαθρομετανάστευσης ε, ή σε αιτήσει ασύλου που δεν έχουν βάση, ε, σε απορριφθήσεις αιτήσει επανειστοχής ή αύξηση ή άμεσο κίνδυνο στην δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ευχαριστώ κύριε Κύρκο. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάιρος Βόλσκι, που είναι εισηγητής ε, για το θέμα αυτό, για το ίδιο θέμα, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγητή για την απελευθέρωση ε, με την Ουκρανία. Το συζητήσαμε χθε. Και κατά τη γνώμη μας, ε, εκφράζουμε την άποψή μας μάλλον για το μηχανισμό αναστολής. Λέμε ότι ο μηχανισμός αναστολής είναι σημαντικό εργαλείο ε, για την εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει μόνο το εσωτερικό στοιχείο, η εσωτερική πτυχή που λαμβάνει υπόψη φυσικά η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά μην ξεχνάμε και τις εξωτερικές, την εξωτερική διάσταση του θέματος πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η ανησυχία που είναι κοινή και για το κοσμοπέδιο και για τη Γεωργία και για την Τουρκία, δηλαδή για όλες αυτές τις συμφωνίες είναι ότι θέλουμε αυτές οι, αυτοί οι όροι στην εξωτερική πολιτική α, απέναντι σε αυτές τις τρεις χώρες να συνεχίσουν να ισχύουν και όχι να υπαναχωρήσουμε όταν δοθεί ε, η απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων στις τρεις αυτές χώρες. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εισάγουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης για να εξασφαλίσουμε ε, την δυνατότητα να επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να ελέγχει ε, εάν εφαρμόζεται η νομοθεσία ε, κατά της διαφθοράς ε, από τις τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Είναι επίσης εργαλείο για την εξωτερική πολιτική και ο μηχανισμός αναστολής της προσπροτείνεται είναι ανεπαρκής. Και κατά γνώμη μας λέμε ότι θεωρούμε ότι αυτός ο μηχανισμός αναστολής προς το παρόν δεν είναι ε, επαρκής γιατί εστιάζει μόνο στους κινδύνους μετανάστευσης και θα πρέπει να συμπληρώσουμε το εξής. Να συνεχίζουν οι χώρες αυτές να πληρούν ε, τα πρότυπα και τα, τους όρους αναφορά στα benchmarks. Όταν δίνεται η απελευθέρωση και εφόσον δεν υπάρχουν μεταναστευτικοί κίνδυνοι, λόγω της απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων κτλ, όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα. Ακόμα και τότε θα πρέπει όμως αυτά τα benchmarks να συνεχίζουν να ισχύουν και να μην αναστέλλονται. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο στη συζήτηση εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο μηχανισμός, ε, αυτό το, το στοιχείο θα πρέπει να προσθεθεί στο μηχανισμό αναστολής. Από τη συζήτηση που είχαμε χθε στην ΑΦΕΤ, εκτιμούμε ότι η πρόταση για να συμπληρωθεί αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, εμείς το υποστηρίζουμε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το μέτρο είναι καθολικό. Δεν αφορά συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Αφορά όλες τις τρίτες χώρες που αποκτούν αυτό το προνόμιο να μην υπόκεινται στην υποχρέωση ε, έκδοσης θεωρήσεων για να μπουν οι υπηκοοί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία, αυτές οι αντικειμενικές προϋποθέσεις να μπουν στη συμφωνία παρόλα αυτά. Η ΑΦΕΤ πιστεύει ότι κάθε συμφωνία κάθε τρίτη χώρα να συμπεριλαμβάνει επίσης και την ε, ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εφόσον το θέλουμε αυτό, με την ίδια λογική, ε, τα δημοκρατικά πρότυπα, ε, οι δημοκρατικές προϋποθέσεις, ε, το κράτος δικαίου κτλ. Όλα αυτά πρέπει να προσθεθούν, ούτω ώστε να συνδέσουμε την ρήτρα αυτή με πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένες προϋποθέσεις χωρίς να αναφέρουμε ονομαστικά κάποιες τρίτες χώρες. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτές τις προϋποθέσεις όπως ε, στις συμφωνίες που συνάπτουμε με τις χώρες ΒΛΑΠ κτλ. Θέλω να σας ευαισθητοποιήσω σε αυτό το θέμα ε, και να σας εκφράσω αυτή την άποψη της ε, ΑΦΕΤ. Ο μηχανισμός λοιπόν αναστολής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους μεταναστευτικούς κινδύνους, αλλά και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δίνουμε αυτό το προνόμιο ε, στις τρίτες χώρες, να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση ούτως ώστε οι στόχοι εξωτερικής πολιτικής να εξακολουθούν να υλοποιούνται και να μην αναστέλλονται. Εν πάση περιπτώσει, να μην υπάρχει υποτίμησή τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Σάριος και ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Αγκώστην για τις τόσο καλά ε, συντεταγμένες τροπολογίες του. που έλαβαν υπόψη τις απόψεις των ε, σκιωδών εισηγητών, διότι ο μηχανισμός αναθεώρησης είναι πολύ σημαντικός ως πρόσθετο εργαλείο για τις διαδικασίες απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τροπολογίες που μιλούν περί ε, κατεξοδοτήτησης πράξεων και την συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Και στην αρχή της διαδικασίας και όταν ξαναβλέπουμε τις θετικές αποφάσεις, μετά από κάποια σπασίματα, πρέπει να θεωρούμε ότι τα κριτήρια, πρέπει μάλλον να φροντίσουμε τα κριτήρια αυτά να είναι σαφή. Και πρέπει να φροντίσουμε και για την ίση μεταχείριση. Όταν υποβλήθηκε η πρόταση αυτή, όπως είπε και ο Σάρις Βόλσκι, ήταν πολύ σημαντικό να λεφτούν αυτές οι διαστάσεις, όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην αξιολόγηση των χωρών και των εθνών για την εφαρμογή όχι του μηχανισμού αναστολής. Rule So at the same time we need to remember about, about... Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε τα δικαιώματα και το σεβασμό τους και το κράτος δικαίου, αλλά και από τη σκοπιά των δικών μας κρατών. Δεν μπορεί λοιπόν να προβλέπουμε αυτές τις προϋποθέσεις και να μην λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια κάτι με το κράτος δικαίου. Και τελευταία παρατήρηση. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε, διότι γνωρίζουμε ότι η απόφαση, μάλλον οι αποφάσεις για την απελευθέρωση θεωρήσεων για την Τουρκία, Ουκρανία, Γεωργία και Κωσυφοπαίδιο, κατά πάσα πιθανότητα θα ληφθούν το φθινόπωρο. Το να αποστείλουμε το μήνυμα προς τους εταίρους μας, κυρίως προς την Ουκρανία και την Γεωργία, ότι εγκρίναμε το μηχανισμό αναστολή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να εργαστούμε αμελητή. Και η τελευταία μου πρόταση, ή δυνατόν, μετά τη λήξη της προθεσμίας της τροπολογίας 22 Ιουνίου, εάν μπορούμε, να επιταχύνουμε λίγο. Και να ψηφίσουμε νωρίτερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. και αν γίνεται να ψηφίσουμε στη Σύνοδο Ολομέλειας του Ιουλίου. Είναι δύσκολο, μεν, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή η ψηφοφορία πριν τις διακοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσεχόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση. Πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές που συνεργάστηκαν. Και να επισημάνω ότι η κύρια ανησυχία μου είναι η εξής έχουμε ένα τρένο εν κινήσει και εμείς μιλούμε για χειρόφρονο συναγερμό. Ίσως πριν αρχίσουμε να μιλούμε για απελευθέρωση από υποχρέωση βίζας, ήταν καλό να εξασφαλίσουμε ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις προκαταβολικά, για να μην χρειάζεται να μιλούμε για χειρόφρονο ασφαλείας. Έχουμε σημαντικό σημαντική αύξηση στον αριθμό επικών τρίτων κρατών ή άλλους παράγοντες κινδύνους, κινδύνου. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε όπως ορίζει και η έκθεση πριν να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός άρσης της διευκόλυνσης. Ωραία κυρίες και κύριοι. Εγώ ρωτάω το εξής λοιπόν. Κοσυφοπέδι, τι θα κάνουμε. Γιατί αν κοιτάξουμε τα δεδομένα από το 2013 μέχρι τώρα, η οι υπήκοοι του κοσμοπεδίου φαίνεται να πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις απειλής και αδικαιολόγητες αιτήσει ασύλου και κίνδυνο απειλής για ορισμένες χώρες συμπεριλαμβανομένες της τσεχικής δημοκρατίας. Το Υπουργείο των Αστερικών, το Μοσπονδιακό ε, της Γερμανίας, μου έδωσε πληροφορίες ότι πολλές φορές ε, παρουσιάζονται στα σύνορα με ε, πλαστά διαβατήρια σερβικά η υπήκοοι του Κοσμοπεδίου, για να μην φαίνεται ακριβώ ότι είναι κόσοβάρι και με, τέτοια διαβατήρια συλλαμβάνονται έχοντα διαπράξει σημαντικά εγκλήματα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Για δε την Τουρκία. Ε, μας ζητήθηκε να επιταχύνουμε τις διαδικασίε ε, ε, άρσης γιατί θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός εκτακτής ανάγκης. <coughs> Ναι, αλλά όταν έχει ένα τρένο εν κίνηση, γιατί εμένα μου συνέβη το να τραβήξει το χειρόφρενο συναγερμού, δεν φέρνει πάντα αποτελέσματα. Καταρχά είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά είναι και επικίνδυνο. Δεν δουλεύει πάντα και δεν δουλεύει αμέσω το χειρόφρενο αυτό συναγερμού. Γι' αυτό λοιπόν, πριν μιλήσουμε για την θεραπεία, πρέπει να μιλήσουμε για την πρόληψη του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή και πάλι, παρακαλώ την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Η κυρία Βαγιαγό Κασίλδο, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Home. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλημέρα σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή, την Επιτροπή σας όλοι για την προτεραιότητα που αποδώσατε σε αυτό το φάκελο και βέβαια την ε, ταχύτατη επεξεργασία του από τον εισηγητή. Αλλά και γενικότερα ευχαριστούμε για τη γενική υποστήριξη που εκφράζει ο εισηγητής και ε, αρκετά μέλη της Επιτροπής σας για την πρόταση αυτή. Ο στόχος της πρότασης ήταν να εξασφαλιστεί η ευελιξία που χρειάζεται ώστε ο μηχανισμός αυτός να γίνει πιο αποτελεσματικός και εύχριστος όποτε Παρίσταται ανάγκη. Λαμβάνουμε υπόψη τι διάφορε τροπολογίε του εισηγητή, την ε, αναφορά, παραδείγματι, στην προσθήκη πρόσθετου κριτηρίου, δηλαδή την ενίσχυση για το, η δημόσια ή την εθνική ασφάλεια ε, κινδύνων για τη δημόσια την εθνική ασφάλεια, τα κατεξοδότης ή κατεξοδότηση πράξης. Ε, η Επιτροπή έχει ζητήσει να γίνει πιο ευέλικτος ο μηχανισμός άρσης εφαρμοστική τράξη, πράξη προβλέπεται αυτή τη στιγμή ε, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση, αλλά βέβαια οι συνομοθέτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν σε ποιο βαθμό θα αξιοποιήσουν τις κατεξουσιοδότες ή εφαρμοστικές ε, πράξεις, δυνάμει της συνθήκης και της ε, νομικής βάσης. Οι στατιστικές που καταγράφονται επίσης στην έκθεση θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικές όπως επισημαίνει και ο εισηγητής. Είναι πολύ σημαντική και σοβαρή απόφαση για τον αποκλεισμό από την απαλλαγή θεώρησης και βέβαια θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Άρα μια τέτοια απόφαση για την άρση της απαλλαγής θα πρέπει να στηρίζεται σε στέρεα αποδεικτικά ε, στοιχεία και δεδομένα και γι' αυτό και εμείς προτείνουμε συγκεκριμένη, μια διατύπωση που αναφέρεται σε ενημέρωση, πληροφορίες και κρυμμένα στοιχεία με βάση τα οποία θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην άρση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Προεδρία. Κέλλη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να σας μιλήσω. Το Συμβούλιο καλωσορίζει το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Δίας Δεμέρα. Μίλησα με κάποιους από τους σκιώδες εισηγητές και μετά από αυτές τις συζητήσεις το Συμβούλιο ε, καλωσορίζει την ε, προτινόμενη μεταρρύθμιση ε, αναστολής του μηχανισμού και το Συμβούλιο ε, πρόσφατα υιοθέτησε τη θέση του για την αναθεώρηση. Ε, το Συμβούλιο θεώρησε, ε, δέχτηκε την πρόταση Κομισιόν και πρόσθεσε και κάποια στοιχεία, ούτω ώστε να λάβει υπόψη τις επιθυμίες των κρατών μελών που θέλουν <clears throat> να ενισχύσουν, να πλουστεύσουν και να ελαστικοποιήσουν το μηχανισμό. Επίσης, Υπάρχει μια σχέση με την ε, δημόσια ασφάλεια και δημόσια τάξη. Και κάποια κράτη-μέλη ακολουθούν έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα κριτήρια, με μια ετήσια έκθεση και αυτόματο μηχανισμό. Εάν μια, η απλή πλειοψηφία των κρατών μελών αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν πληρεί τα κριτήρια, τότε το μέτρο θα πρέπει ε, να εφαρμοστεί για μια προσωρινή αναστολή 6 μηνών. Κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο πιστεύουν ότι η θέση σε ισχύ του μηχανισμού είναι προϋπόθεση για την απελευθέρωση, ε, την υποχρέωση θεωρήσεων για την Τουρκία, Γεωργία, Ουκρανία και Κωσυφοπαίδιο. Και για να μπορέσει να εγκρίνει την απελευθέρωση, το και να εγκρίνει μάλλον την αναθεώρηση του μηχανισμού, περιμένουμε τη θέση του Κοινοβουλίου και ένα σύντομο τρίλογο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα, τελευταίος ο κύριος Ντίας Δεμέρα, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα νέες παρεμβάσεις και πολλές παρεμβάσεις που σας δείχνουν πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ όλους για όλες τις ιδέες. Θα ξεκινήσω με την ε, κυρία Ιώτοβα. Ευχαριστώ κυρία μου για τα λόγια σας. Άκουσα με πραγματικό ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Και αυτό που είπατε για το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και εσείς και εγώ ξέρετε ότι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, στο ίδιο τρένο βρισκόμαστε, το τρένο αυτό πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα ίδια πρεσβεύουμε. Επίσης, χαίρομαι που τονίσατε τη σημασία ε, με έμφαση των ε, κατεξοδότηση πράξεων, ε, όπου αναδεικνύεται η εξουσία ως συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιβεβαιώνεται με την ομολογία του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου. Ο επόμενος ε, ομιλητής έφυγε και δεν θα του απευθύνω κάποια σχόλια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι που στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν. Η κυρία Βιόρ μίλησε εξ ονόματος της ε, Κριστίν. Και με σας ε, συμφωνώ ή με την Κριστίν. Όντως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις κατεξιοδότηση πράξεις. Σας ανησυχεί και σας και εμένα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των, στις τρίτες χώρες. Να σας πω Κοιτάξτε ε, τι λέω στο σημείο 3, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ε, υπηκών τρίτων χωρών. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Άρα συμφωνούμε απόλυτα. Ο κύριος Μπόνι, ο αγαπητός μου φίλος, με πολύ αδερφικό τρόπο με χαιρέτησε την προσπάθειά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας με τη σειρά μου. Χαίρομαι λοιπόν επίσης που στηρίζετε τη θέση μου για τις κατεξιοδότηση πράξης που δίνει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο, που δίνουν μάλλον οι πράξεις αυτές πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με ισοτιμία με το Συμβούλιο. Συμφωνώ για αυτό που είπατε για τη Γεωργία και την Ουκρανία ε, απόλυτα. Και συμφωνώ και, τα, και με τα όσα είπατε για την Τουρκία. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να κινηθούμε ε, πιο γρήγορα. Μ' άρεσε που το άκουσα, μακάρι. Ε, πριν από μία εβδομάδα με υποδείξατε ως ε, εισηγητή. Ευχαριστώ και το φίλο μου τον Τόμας για τα πολύ συμπαθητικά του λόγια. Μου άρεσε πολύ αυτό, αυτή η εικόνα έτσι με το φρένο και το τρένο ας πούμε που χρησιμοποίησατε. Θα πρέπει έτσι να διαφημίσουμε αυτό το μηχανισμό ως ένα ε, φρένο που το πατάμε όταν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά που είπατε για το κοσμοπέδιο τα λαμβάνω υπόψη επίσης ε, υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει πρόβλημα με τις κακέ στατιστικέ προφανώς. Και για το θέμα της Τουρκίας, προφανώς, είναι ανησυχητικό θέμα, δεν το συζητώ. Και πρέπει να τη συνδέσουμε αυτή την πρόταση για την Τουρκία με το φρένο αυτό που είπαμε. Ευχαριστώ την Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που με πολύ διπλωματικότητα έλαβε υπόψη τις τροπολογίες και να σας υπενθυμίσω, Κομισιόν, ότι στις θέσεις σας, ε, όπου αναφέρεται η χρήση των κατεξιοδότηση πράξεων, αυτές οι προτάσεις ακριβώς ε, απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 16 Ιουλίου πέρυσι. Επίσης, η Επίτροπος Σεσίλια Μάλστρομ σας είχε πει ε, ότι θα έπρεπε ουσιαστικά να μην προσφύγετε με αυτή τη θέση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν το κάνατε. Επίσης, καταλαβαίνω ότι οι στατιστικές έχουν τεράστια σημασία. Τώρα, για την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, έχω ήδη συνεργαστεί μαζί της και εκτιμώ την επαγγελματικότητά της. Θέλω να το πω πραγματικά, έτσι, φωναχτά αυτό, να το ακούσουν όλοι. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την το μηχανισμό να τον καταστήσουμε πιο ελαστικό επίσης, το μηχανισμό αναστολή. Το θέμα της δημόσιας ασφάλεια προφανώς μας ενδιαφέρει. Προφανώς και θα πρέπει να έχουμε ένα εύκολο και γρήγορο εργαλείο για να τιμωρήσουμε τους παραβάτες, δηλαδή τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν σέβονται τους κανόνες. Σας ευχαριστώ όλου για τι προτάσει, σα. Θα συνεχίσουμε τι εργασίε μα με την ταχύτητα που εσείς θα μας επιτρέψετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντίας Δεμέρα. Η προθεσμία για την υποβολή των πολεμιών είναι 22 Ιουνίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην ΛΥΜΠΕ προβλέπεται στις... Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Α, κάτι ξέχασα. Ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά που είπε ο κύριος ε, Σάριος Βόλσκι. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα. Σας είχα αφήσει για το τέλος θα λάβουμε πραγματικά υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη σημασία που έχει η αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής και οι επιπτώσεις της αναθεώρησης αυτής στην εξωτερική πολιτική. Ε, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και συγγνώμη που δεν σας ανέφερα πριν. Σας είχα αφήσει για το τέλος για να δώσω έμφαση στα όσα είπατε. Ευχαριστώ κύριε Αντίρευτε Μέρα. 22 Ιουνίου μεσημέρι, τελική προθεσμία, 12 Ιουλίου η ψηφοφορία στη Λίμπε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στην όλη συζήτηση και τώρα στρεφόμαστε στο επόμενο σημείο, στην ημερήσια διάταξη, σημείο 7. Στι 7 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για το λεγόμενο Σύμφωνο Μετανάστευση. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και πώς σκοπεύει να την αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Λεωνέλο Γκαμπρίτσι, διευθυντή ε, για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης συμπεριλαμβανόμενης της μετανάστευσης από την ΕΕ που θα μας παρουσιάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θα έχουμε και συμμετέχοντες από τις Επιτροπές ΑΦΕΠ, και ΔΕΒΕ για να έχουμε διάλογο για το θέμα αυτό. Κύριε Γκαμπρίτς, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρεμπιπτόντως, είπατε ότι προσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είμαι από την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Όμως αγαπώ ακόμη την Επιτροπή, γιατί από εκεί προήλθα. Και πηγαίνουμε έτσι κι χερι χέρι-χέρι μαζί. Να πω ότι θα έχετε δει, ελπίζω όλοι, την ανακοίνωση αυτή καθεαυτή και θα έχετε λάβει και όλα τα δημοσιεύματα στον τύπο που τη συνοδεύουν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι στο τέλος υπάρχει μια σύσταση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να την υποστηρίξει. Οπότε το επόμενο βήμα, το πλέον σημαντικό, είναι να βεβαιωθούμε ότι η αρχική κάτω των κυβερνήσεων θα υποστηρίξουν την ε, έκθεση αυτή, την ανακοίνωση αυτή και τις ε, προτάσεις της. Αυτό που είναι καθοριστική σημασίας ως προς την ε, απαρίθμηση μηνυμάτων στην ανακοίνωση αυτή είναι μια δίπτυχη προτεραιότητα. Πρώτα απ' όλα να επαναληφθούν κάποιες αρχές και προτεραιότητες που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα. Θέλουμε να επαναληφθούν και να ακουστούν, να εγκριθούν από τους αρχηγούς και των κυβερνήσεων η αρχή της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης σε πρώτη φάση και δεύτερον να ανοίξουμε το δρόμο για ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στον τομέα αυτό, στην εξωτερική διάσταση, που να καλεί και τα κράτη-μέλη να αρχίσουν επιτέλους να συμμετέχουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Λίγα σύντομα λόγια για αυτές τις δύο πτυχές. Για τις αρχές λοιπόν που θέλουν να ξανακουστούν από αυτήν την ανακοίνωση, η πρώτη είναι θεμελιώδης. Ό,τι και αν κάνουμε στην εξωτερική διάσταση, οι τρίτες χώρες θα πρέπει να μαζί, μαζί μας σε σχέση εταιρική. Τι θα πει αυτό. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε το μήνυμά μας. Αυστηρός στο θέμα των επιστροφών. Η προηγούμενη συζήτηση για τη μετανάστευση που είχε περάσει και στα χέρια των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη, που σωστά είχαν επικεντρωθεί στα ζητήματα αυτά, είχε ασχοληθεί πιο πολύ με αυτή τη διάσταση. Δεν μπορούμε όμω να λέμε σε τέτοιε χώρε μόνο ότι θα σα δίνουμε κάρτε, ε, αν θα σα δίνουμε καρότα εάν ε, πάρετε πίσω κάποιου ανθρώπου, ενώ θα σα δώσουμε ε, μπαστούνια εάν ε, δεν το κάνετε. Το ζητούμενο είναι πώς θα βοηθήσουμε τις χώρες αυτές, πώς θα καταφέρουμε χώρες αυτές να μας βοηθήσουν γενικώ με το πρόβλημα της μετανάστευσης. Πολλές φορές και οι ίδιες γνωρίζουν φοβερές πιέσεις λόγω της μετανάστευσης, όπως η Τινησία. Θα έπρεπε και δικαίω να συζητήσουμε με τους Τινήσιους για το πώς να κάνουν εκείνη μια προσπάθεια για τις επιστροφές για να αποδεχτούν αυτού που του επιστρέφουμε, του λαθρομετανάστε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και εκείνοι έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο, ίσω και παραπάνω, ε, εκτοπισμένου που έρχονται από την Λιβύη. Συντομεύω κάπω, αλλά το πρώτο μήνυμα είναι ότι αυτό που θα συζητάμε με τι τρίτε χώρε δεν είναι απλώ η διάσταση των δικών μα των συμφερόντων. Πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τι μεταναστευτικέ ροέ και βάση του υπάρχοντος πολιτικού διαλόγου. Το δεύτερο στοιχείο που επαναλαμβάνεται στην ανακοίνωση είναι ακριβώς αυτή η ολιστική προσέγγιση. Όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργοποιηθούν στην διάρθρωση του πολιτικού μας διαλόγου. Τι εννοώ άραγε. Ε, να πάρω πάλι το παράδειγμα της Τινησίας που είναι μέρος της πολιτικής γειτονίας. Υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής, υπάρχει πρόγραμμα δράσης, είναι περιοχή ελεύθερου εμπορίου για τα αγαθά που παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τους ρωτήσετε τι μπορούν να κάνουν όχι μόνο συγκεκριμένα αλλά γενικώ για να αντιμετωπίσουν τα μεταναστευτικά προβλήματα βρίσκεται μπροστά σας αυτή την πλατφόρμα ήδη υπάρχει Συζητάμε το εμπόριο, τη γεωργία, την ασφάλεια, το κράτος δικαίου. 360 μοιρών ολιστικό διάλογο έχουμε μαζί τους. Εάν δείτε ότι στο διάλογό μας υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να τα, να τα ε, επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου χάρη στη συμφωνία Κόπεν ε, με την Τινησία όπου μπορούν εταιρείε χαμηλού κόστους να δραστηριοποιηθούν στην Τινησία αυτό γίνεται αποδεκτό και προκύπτει από τις κοινοτικέ ε, αρμοδιότητες λόγω των ανοιχτών ουρανών του συστήματος Open Sky λόγου χάρη. Αλλά είδαμε ότι αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει αν θέλουμε να πάμε παραπέρα στη συνεργασία μας. Οπότε στην ανακοίνωση δηλώνατε σαφώ ότι τα κράτη-μέλη τα ίδια πρέπει να βάλουν πόδι. Έχουν ιστορικούς δεσμούς και σχέσεις με κάποιες από αυτές τις χώρες. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης που έχουν ε, πληγεί ποια μέσα την μετανάστευση από κάποιες τέτοιες χώρες, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λυθούν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας μόνο τις γαλάζιε σημαίες στο Open Sky. Πρέπει να υπάρχουν και διμερείς πρωτοβουλίες. Προσπαθώ να τα πω σύντομα και γι' αυτό ένα κεφαλαίο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα θέματα τη μετανάστευση για να μπορέσουμε το πνεύμα της Λισαβόνας να το κάνουμε πραγματικότητα. Και το τρίτο, το τρίτο μέρος της ανακοίνωσης, που είναι κάτι θεμελιώδες και για την ανακοίνωση, εάν κάτι θέλουμε να πετύχουμε, είναι ολιστική προσέγγιση, εταιρική σχέση και καταδικασμένη να δουλεύουμε μαζί ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κράτη-μέλη σε πλήρη ε, παραλληλισμό. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μετανάστευση. Αυτό αναφέρεται και ως, ε, είναι γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με την κλασική μα αναπτυξιακή βοήθεια, τα γνωστά κονδύλια. Ακόμη και τα κρατημέλη κάνουν προσπάθειε να βρουν επιπλέον χρήμα για την κλασική αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό δεν θα αρκέσει. Δεν θα αρκέσει για να αντιμετωπίσουμε τι μεσοπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε απειλέ από τι χώρε αυτέ. Διότι η τάση είναι οι χώρε αυτέ, τουλάχιστον κάποιε από αυτέ, και όλο ιδιαίτερα στην Εποσαχάρια, Αφρική και την Ασία, είναι να γίνονται όλο και φτωχότερε, να παράγουν δηλαδή φτώχεια, άρα και όλο και περισσότερου ε, μετατοπιζόμενου, εκτοπιζόμενου ε, ανθρώπου. Χρειάζεται μια απόκριση από τη διεθνή κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βοηθήσουμε και να έχουμε κοινωνικο-οικονομικές βιώσιμες λύσεις και να είναι και αυτοί κοινωνικο-οικονομικοί μας εταίροι που να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα της κυριαρχίας τους για τη διαχείριση των σύνορων και το καθεξής του το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν η λογική του προγράμματος επενδύσεων δεν έχει να κάνει μόνο με την προσφορά χρήματος είναι η προσφορά κινήτρων για επενδύσεις. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετάσχουν. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και ιδίως στην Αφρική. σε σχέση με την Κίνα έχουμε χάσει κάπως έδαφος. Μεσοπρόθεσμα λοιπόν και μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η στρατηγική μας θεώρηση για τις εταιρικές μας σχέσεις και από κοινωνικονομικής σκοπιάς με τις χώρες αυτές. Αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε ακόμη περισσότερο βέβαια. Όμως είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε τις τάσεις που δείχνουν ότι Μπορεί να πάνε χειρότερα τα πράγματα. εάν δεν ε, βοηθήσουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 100-300.000 ε, άτομα, 2 3 εκατομμύρια πρόσφυγες ε, μπορεί να έρθουν ε, στο επόμενο διάστημα στην Ευρώπη, αυτό ακούμε, αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι στον πλανήτη υπάρχουν 60-80 εκατομμύρια εκτοπισμένοι ε, ανά τον πλανήτη. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρωταγωνίστριας στη διεθνή κοινότητα είναι να συμπαρασύρει σε αυτή την προσπάθεια τη διεθνή κοινότητα. Και στη σύνοδο του ΙΕ τον Σεπτέμβριο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και με την πρωτοβουλία του Προέδρου Ομπάμα για τους πρόσφυγες. Με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστούμε κύριε Καπρίτσι. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Κουτσέκεβιτ. Ζητώ συγγνώμη για την, προ... για την προφορά. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμπληρώσω στα όσα είπε μόλις ο συνάδελφος από την ε, και δεδομένου ότι η ανακοίνωση είναι κοινή ανακοίνωση Επιτροπή και της Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Για τη Γενική Διεύθυνση λοιπόν των Εσωτερικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ανάπτυξη των εξή αξιών, συνέχεια αφενός δράσεων, καταγραφεί ως εκ τούτου πρώτα του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα εξωτερικά αλλά και εσωτερικά γιατί έχουμε αναπτύξει διάφορες προσεγγίσεις προς τις τρίτες χώρες όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν πάντα οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις. Γι' αυτό και βρισκόμαστε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αλλά πάντως δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για την ε, μεταναστευτική κινητικότητα. Έχουμε προσπαθήσει να οργανώσουμε διαφορές δέσμες σε σχέση με κινητικότητα, θεωρήσεις, ούτω καθεξής, εταιρικές σχέσεις κινητικότητας ε, και θεωρήσεων και βεβαίως ε, διάλογος ψηλού επίπεδου που οργανώθηκε τους τελευταίους μήνες, σύνοδος της Βαλέτα, όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή με βάση τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε προς μια πιο αποτελεσματική οργάνωση. Εξού και το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης εστιάζεται στην ιδέα των μεταναστευτικών εταιρικών σχέσεων. Αυτές είναι το σημαντικότερο κομμάτι που θα μας επιτρέψει μετανάστευση ε, να θέσουμε τη μετανάστευση στο επίκεντρο των εξωτερικών μας σχέσεων. Μέχρι τώρα είχαμε τα εργαλεία της Γενικής Διεύθυνσης των Ιστορικών στην ενίσχυση των σχέσεων με τις τρίτες χώρες. Με την ανακοίνωση της Επιτροπής προφανώς και ξεκάθαρα προάγεται μια προσέγγιση ευρύτερη, ολιστική, αναπτύσσεται δηλαδή μια προσέγγιση με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων. Και εδώ μιλούμε για εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες, μια κοινή επιχείρηση σε βάση κοινή ευθύνη, συνυπευθυνότητα. Αυτή είναι η επιλογή μα και περιμένουμε βεβαίω μετά τις ξεκαθαριστικές μας δεσμεύσει και αντίστοιχε δεσμεύσει από πλευρά των τριτών κρατών. Επίσης, πολύ σημαντικό, είναι και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στην υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί να αποτελέσει ένα εγχείρημα μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια της σημασίας των θεμάτων που διακυβεύονται, αλλά και της σημασίας των σχέσεων με τις τρίτες αυτές χώρες. Ορισμένα κράτη-μέλη Φερρυπίν μπορεί να έχουν και προνομιακές σχέσεις μαζί τους, που δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, ας δείξουμε μια συνοχή και ας μιλήσουμε την ίδια φωνή. Πέρα λοιπόν της ε, συνιστώσας της ε, μετανάστευσης υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις που θα θέλαμε από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης των Εσωτερικών να επισημάνουμε, θέματα δηλαδή εμπορίου, αναπτυξιακής βοήθειας ή άλλα τομεακά θέματα σημασίας για την τρίτη χώρα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συζήτηση. Βεβαίως και θα πρέπει να ακούσουμε τι θέλει αυτή η τρίτη χώρα, τι περιμένει, τι συμφέροντα έχει. Βραχυπρόθεσμα έχουμε τρεις στόχους ορίσει ε, για τις εταιρικέ σχέσεις, να σώζονται ανθρώπινες ζωές, να λειτουργήσει το σύστημα της συνεργασίας της επιστροφές και η ανθεκτικότητα των τρίτων κρατών που είναι κυρίως χώρες διέλευσης ή υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών ή προσφύγων, οι ίδιες, να υποστηριχθεί. Μακροπρόθεσμα βέβαια πρέπει να καταπολεμηθούν οι ρίζες της ε, μετανάστευσης. Οικονομική διάσταση επίσης. Έχει αυτή μεγάλη σημασία, αν και από πλευράς μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η ανάπτυξη έχει να δώσει πολλά σε οικονομική ενίσχυση, αλλά εμείς ως Γενική Διεύθυνση Ιστορικών μπορούμε να ενθαρρύνουμε προς ε, διάφορες κατευθύνσεις, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την ανακοίνωση, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα γεωγραφική διάδοση, διάχυση. Ορίζουμε κάποιες χώρες προτεραιότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρετούμεθα από την συνεργασία ε, με άλλες τρίτες χώρες που δεν αναφέρονται ρητά. Απλώς εστιζόμαστε περισσότερο στις τρίτες χώρες που αναφέρουμε και κυρίως τις οδούς της κεντρικής Μεσογείου, εξού και αναφέρονται οι πέντε ε, χώρες που βλέπετε χώρες διέλευσης και προέλευσης για, τις, ε, για, την, κεντρική, ε, για την οδό της κεντρικής Μεσογείου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αγνοούμε τη σημασία άλλων τρίτων χωρών ή ότι εγκαταλείπουμε συνεργασίες που έχουμε ήδη αναπτύξει. Όλα αυτά σε συνεργασία και με την κυρία Μογκερίνη και τις υπηρεσίες της για να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός ώστε να εξετάσουμε εσωτερικά πώς μπορούμε να οργανωθούμε να δώσουμε ε, σάρκα και ουστά σε, αυτή την, ε, σε αυτό το εγχείρημα να δούνε και τα κράτη-μέλη πώς θέλουν να το χειριστούν και βέβαια στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή με τις τρίτες χώρες το πνεύμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συζήτηση. Λαουριστίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για την ε, πρακτική υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Τι είδους ε, επιτήρηση προβλέπετε να εγκαθιδρυθεί και πώς θα ενημερωνόμαστε. γιατί από χτε με κάποιες επαφές που είχα με προσώπους δημοκρατικών δυνάμεων της Τουρκίας ακούσα πολύ, μεγάλη, πολύ ανησυχητικές ε, ε, τοποθετήσεις για το κίνδυνο τα χρήματα που διτίθεται στην Τουρκία να πάνε στα λάθος χέρια και σε λάθος χρήση. Επίσης τεχνική ενίσχυση, τι μπορεί να σημαίνει. Πάντα βλέπουμε σε κάθε έκθεση και για κάθε γωνιά του κόσμου να ζητείτε τεχνική υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα τμήμα τεχνογνωσίας, υπάρχει ένα τμήμα, τμήμα ανθρώπινων πόρων. Πρακτικά τι σημαίνει. Ευχαριστώ, Μπιόρκ. Ευχαριστώ. Όπως και με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων, έχουμε την εντύπωση ότι το μόνο που θέλουμε όλοι είναι να σταματήσουμε του πρόσφυγες από το να μπαίνουν στην Ευρώπη. Ότι είναι ο μόνος φόβος μας, το μόνο μέλημά μας. Ε, όπως ε, σε αυτό το σύμφωνο με την Τουρκία είναι σαν να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής για να σταματήσουμε τους μετανάστες. Ε, την, αναπτυξιακή πολιτική, την εμπορική πολιτική, όλες τις πολιτικές. Και αυτή η πρόταση λοιπόν είναι πονίδιστη για αυτό το λόγο. Αντίθετα, καλό είναι να έχουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν προτείνουμε πραγματικές συμφωνίες. Στην πραγματικότητα περί πρόκειται. Ε, έχουμε δικτατορικά καθεστώτα, ε, καταπιεστικά καθεστώτα ε, στο Σουδάν, στην Ερυθρέα κτλ. Και κάνουμε outsourcing του ελέγχου των συνόρων μας, στην πραγματικότητα στις χώρες αυτές. Αναθέτουμε σε αυτές τις χώρες την ευθύνη. Θε, ορισμένοι είπαν μάλιστα, ορισμένοι πολιτικές δυνάμεις, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, σε διάφορα νησιά, ας πούμε, ε, κλειστούς χώρους για να στηβάξουμε εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Στην πραγματικότητα, ε, παίζουμε το παιχνίδι ε, καθεστώτων χωρών που πραγματικά θέλουν να καταπιέσουν. Φαντάζομαι ότι στην Ολομέλεια πολλές πολιτικές ομάδες θα εκφράσουν ε, επικριτική ε, άποψη για τη θέση αυτή. Στην πραγματικότητα θέλουμε λύσει με αλληλεγγύη, ούτω ώστε να παραμείνει ανοιχτό χώρο η Ευρώπη και να καλωσορίσουμε τους μετανάστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, θα, ότι ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο ε, για την Αφρική με, μεγάλο, με μεγάλα σχέδια συνεργασία ε, είναι κάτι το πολύ θετικό. Όμω, ανησυχώ διαβάζοντα αυτή την πρόταση. Καταρχάς επικεντρώνει στο να αυξήσει την ε, συνεργασία με τρίτες χώρες, ούτως ώστε να εμποδίσουν ουσιαστικά τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη φτώχεια και τον ε, πόλεμο να μετακινηθούν προς την ε, Ευρώπη. Το, τις σχέσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες να τις βασίσουμε σε κάτι τέτοιο, ας πούμε, σε αυτή την προϋπόθεση, νομίζω ότι προδίδουμε τις σχέσεις. Γιατί στην πραγματικότητα ε, επικεντρώνουμε ε, στην, των συνόρων. Δεν, αυτό δεν δημιουργεί ούτε ευκαιρίες, ούτε μειώνει τις, αν, ανισότητες, ούτε λύνει τα προβλήματα. Νομίζω ότι παίρνουμε, παίρνουμε λεφτά από την αναπτυξιακή συνεργασία και τα δίνουμε ε, στο, στη διαχείριση των συνόρων και, στο, και στην οικοδόμηση δυναμικού σε αυτές τις χώρες για να διαχειρίζονται τα σύνορά τους. Στην πραγματικότητα εξωτε, ε, αναθέτουμε στο εξωτερικό ας πούμε τις δικές μας ευθύνες ε, και το θέμα των συνόρων μας. Εάν τα κράτη-μέλη είχαν ήδη ενεργοποιήσει τις κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις ε, στα, πάνω στα οποία δεσμεύτηκαν πέρυσι, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πρόεδρε ίσως έχει νόημα. Να σας πω ότι παρίσταμαι εδώ γιατί είμαι ο εισηγητής για τη μόνιμη αναπτυξική βοήθεια στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Και επομένως ερμηνεύω κάποιες από τις, τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανάπτυξης πάνω σε αυτή την πρόταση. Και τη συνδέω με, τις, ε, με τις ε, επικρίσεις που ακούσατε από τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Καταρχάς, ε, το θέμα της μετανάστευσης το βάζουμε στο κέντρο της ε, ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης. Επιτέλους, συνειδητοποιούμε ότι η Αφρική είναι ένα από τα εξωτερικά μας σύνορα στην πραγματικότητα. Και με πολιτικό αλλά και με γεωστρατηγικό τρόπο είναι στη γειτονία μας η Αφρική. Και ή θα λύσουμε τα προβλήματα φτώχειας και τα προβλήματα ε, σειράξεων ή αλλιώς θα έχουμε μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική ροή από, από την Ήπειρο αυτή προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Και θα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που θα φεύγουν λόγω φτώχειας ή πολέμου. Επομένως, να θέσουμε το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων στο πλαίσιο της εξωτερικής μας δράσης μου φαίνεται ότι είναι εκ των όνων Δεύτερον, η εστίαση στην εταιρική σχέση είναι η μόνη δυνατή εστίαση που μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας μονομερός να επιβάλλουμε μια συγκεκριμένη πολιτική στις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε συνεργασία σε εταιρική σχέση μαζί τους. Οι ανησυχίες προέρχονται από διάφορους ε, τομείς και για διάφορους λόγους. Όπως υπόθηκε καταρχήν είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την πολιτική ανάπτυξη μόνο επιβάλλοντας όρους και προϋποθέσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία προϋπόθεση και να μην βάζουμε κανέναν όρο στις τρίτες χώρες. Φυσικά όμως η πολιτική ανάπτυξη πριν από οποιαδήποτε νέα πρόταση, ε, πριν από οποιαδήποτε αναθεώρηση, έχει προϋποθέσεις. Δηλαδή, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλή διακυβέρνηση. Συνδέεται και με άλλες προϋποθέσεις, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται με την πολιτική θέση που μπορεί να πάρουν οι χώρες αυτές που λαμβάνουν αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί ο στόχο τη αναπτυξιακή πολιτική είναι η καταπολέμηση τη φτώχεια και η δημιουργία ευκαιριών ζωή. πολύ λιγότερο για την, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν μπορούμε να βάλουμε προϋποθέσεις. Φυσικά υπάρχουν διάφορες αρχές. Μεταξύ αυτών είναι προφανώς η ουδετερότητα και η αμεροληψία που είναι, υποτίθεται αρχέ, που είναι προφανώς αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με οποιασδήποτε προϋποθέσεις που επιβάλλονται άνωθεν, ας πούμε. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στο, στη δημοσιονοπτική πτυχή αυτού του θέματος. Ας μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι. Αυτό που έχουμε είναι, συσσωρεύουμε πόρους που προβλεπόταν στο σχέδιο για τη Συρία, προέρχονται από το Ταμείο Ανάπτυξης και ούτως ή άλλως είναι πολύ περιορισμένοι. Αν λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση του προβλήματος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι σωστό, ε, καλό είναι που ακούσαμε ότι η Κομισιόν ε, το φθινόπωρο θα έρθει με μία πρόταση που για επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να βάλουν τα κράτη-μέλη το χέρι στην τσέπη, κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόταση, ε, υποτίθεται, ας πούμε, αυτά τα 72 δισεκατομμύρια, έτσι, τα μισά πρέπει να τα βάλουν τα κράτη-μέλη. Στην πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψη μας τι συνέβη την τελευταία χρονιά, ε, τα πράγματα δεν είναι πολύ ρόδινα. Η Αφρική είναι μια τεράστια ήπειρο. Και αν δεν κάνουμε μια αντίστοιχη προσπάθεια με τα 72 δίσενο, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστούμε σωστά αυτά τα σύνορα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επαρκή προπολογισμό. Έτσι. Δεν έχει επαρκή πόρους. Ε, αυτό το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εκτός, ε, πέρα από αυτή την έκθεση, δηλαδή πέρα από αυτή την επιτροπή. Εάν δεν ε, λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης, δεν φτάνουμε πουθενά. Ο κ. Κυρικόπου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προτάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, το ίδιο και τα σχόλια της Επιτροπής. Αλλά αυτό που θα ήθελα εγώ να σχολιάσω είναι το θέμα των κονδυλίων και ο τρόπος που χρησιμοποιείται ο όρος επιδόσεις. Όταν ε, μιλάμε για μετανάστευση είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε τέτοιους όρους και έννοιες. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των επιδόσεων σε σχέση με, τις, τα με τη μετανάστευση και το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Το πώς δαπανώνται σε, σε λεπτομέρειες έτσι όπως προτείνονται. Θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα λοιπόν. Εάν θυμηθούμε αν θυμηθώ μάλλον τη δική μου εμπειρία ως Υπουργού Μετανάστευσης στη δεκαετία του 90, δεν ήταν τόσο εύκολο να ξεχωρίσουμε τις θετικέ από τις αρνητικέ εμπειρίε και σίγουρα υπάρχουν κάποιε χώρε εξίεπινες που θέλουν να συνεργαστούν, αλλά χρησιμοποιούμε εδώ και του όρου επιπτώσει για αυτούς που αρνούνται. Αυτό, αυτό πραγματικά μου θυμίζει το τι συνέβαινε στην περίπτωση που ήμουν μέλος τη κυβέρνηση και υπήρχαν επιπτώσει εντό εισαγωγικών για όσου δεν ήταν αρκετά πιστή στην κυβέρνηση. Τέλο πάντων, τα σχόλια έχουν να κάνουν με την εσωτερική μα πολιτική, αλλά με ενδιαφέρει και η άμεση σχέση μεταξύ τη ε, νόμιμη μετανάστευση και το πώ αυτή αντιμετωπίζεται σε σχέση με την παράτυπη. Μα λέγεται πάντοτε ότι αν αυξηθούν οι ευκαιρίε για νόμιμου μετανάστε, αυτό από μόνο του θα μειώσει την πίεση τη λάθρο μετανάστευση ή τη παράτυπη. Δεν είμαι βέβαιο. Θα ήθελα να έχετε περισσότερα στοιχεία αριθμητικά για το τι πραγματικά συμβαίνει. Διότι έχω κάποιε αμφιβολίε. Και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ό,τι άλλο και αν προβλέψουμε, το βασικό είναι να έχουμε απόλυτη σαφήνεια στην προσέγγιση μα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ανταμοιβέ επιπτώσει, για νόμιμη παράτυπη μετανάστευση, για ειδοποίηση των κρατών και των ατόμων, για τι περιστάσει, του όρου, ε, υπό του οποίου μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει. Εδώ πρέπει να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια. Κάποιες φορές διερωτώ με μήπω χανόμαστε πάλι σε ένα κείμενο από πολλά ωραία λόγια ενώ στην πραγματικότητα η πράξη είναι τελείω διαφορετική. Ευχαριστούμε κύριε και κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικό όταν ακούω τον Τίμωθη Κύρκοπ πάντοτε αισθάνομαι ότι εμπνέομαι. Όχι απλώς έχει πάντοτε πολύ πνεύμα και χιούμορ, και τα φέρνει αυτά εδώ στη συζήτηση, αλλά έχει και πολύ φαντασία και δημιουργικότητα. Ε, κάτι που είναι χρήσιμο για όλους μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση, να σκεφτούμε το πλαίσιο εντό του οποίου υποβάλλεται. Το πλαίσιο είναι το εξή. Έχει πάρει φωτιά ο κόσμος γύρω μας. Βεβαίως πάντοτε πρέπει να συνεργαζόμαστε και να έχουμε εταιρικέ σχέσεις, εταιρικέ σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, αλλά το ερώτημα είναι σε τι βαθμό μήπως δεν έχουμε ακόμη καταλάβει πώς πρέπει να ε, διαχειριστούμε τα σύνορά μας, πώς μπορούμε να εκχωρήσουμε τις ανθρωπιστικές μας ευθύνες. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ξανακάνουμε μια να αναλάβουμε τη συμφωνία με την ε, Τουρκία ε, σε χώρες όπως η Λιβύη. Το είπε σήμερα ο Αυστριακός Υπουργός ο νέο Υπουργό για τι Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Πριν από 10 μέρες τοποθετήθηκε για την απόλυτη ανάγκη του να ε, κάνουμε συμφωνία με τη Λιβύη. Μα είναι κράτος αποτυχημένο η Λιβύη. Ε, θα προχωρήσουμε μετά την Τουρκία και στη Λιβύη και ποια θα είναι η επόμενη και μεθεπόμενη χώρα. Αυτά λίγο να τα σκεφτούμε και ιδίω ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Ήδη δαπανούμε πάρα πολλά με την δήλωση αυτή με την Τουρκία. Περισσότερα χρήματα από όσα δαπανούμε για την αναπτυξιακή μας βοήθεια για τον υπόλοιπο κόσμο, από ό,τι για τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι πάρα πολύ το χρήμα. Τι να κάνουμε λοιπόν εδώ, τι απομένει, ποιο θα είναι το περιεχόμενο, το πλαίσιο εντό του οποίου θα δράσουμε και θα ενεργήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. την έννοια της Ευρώπης του οχυρού αυτού θα την εφαρμόσουμε καθόλου. Πολύ φοβάμαι ότι η πρόταση αυτή θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά ακριβώς σε αυτή την περιφρουρούμενη την Ευρώπη. Και αυτό πάρα πολύ με ανησυχεί. Πάντοτε πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις γειτονικές χώρες. Αλλά το να, αναθέσουμε εξωτερικώ αυτά τα θέματα, όπω τη διαχείριση συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το βρίσκω παράδεκτο. ευχαριστώ πολύ, κυρία Χόλμαγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το μείγμα αυτών των παρατηρήσεων που ακούστηκαν, που δεν έχουν πάντα άμεση συνάφεια με το θέμα που συζητούμε, αν και βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε και με ε, δεσμεύσεις αναπτυξιακές της ε, Ένωσης ε, σε τρίτες χώρες. Θέλω ωστόσο να πω ότι πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο και αναφερόμενοι προς τους ε, συναδέλφους σοσιαλιστών ε, δημοκρατών θα επισημάνω πως οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές φεύγουν από τις χώρες τους λόγω της ε, κατάστασης που αντιμετωπίσουν γιατί δεν υπάρχει οργανωμένη κρατική δομή, δεν υπάρχει αστυνομία που να τους προστατεύει, δεν έχουν μέλλον προοπτικές. Και άρα πρέπει να επενδύσουμε και στις χώρες αυτές. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι να φεύγουν ως το δυνατόν περισσότεροι από τις χώρες τους για να τους υποδεχόμαστε εμείς, αλλά να τους δίνουμε προοπτικές να μένουν εκεί. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ και την προσέγγιση της Επιτροπής. Και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ανθρωπιστική ενίσχυση και ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση των περιοχών και χωρών της Αφρικανικής Υπήρου που το έχουν ανάγκη. Αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο κρατών μελών να εκδηλώνεται. Και από την άλλη, αν καταλαβαίνω καλά τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σκοπεύει ε, να οικοδομήσει ένα νέο ευρωπαϊκό φρούριο, την Ευρώπη ως φρούριο, αλλά αντιθέτως ε, να αντιμετωπίσει και να οργανώσει κατά κάποιο τρόπο ροές τις οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν τα κράτη μόνα τους γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιπαραθέσεις και δυσκολίες επειδή ακριβώς τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να συνεννοηθούν και να βρουν λύσεις οι οποίες να είναι αποδεκτές και για τους πολίτες τους. Ε, υπερβολικές λοιπόν ροές ή η υποδοχή των γνησίων προσφύγων είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις που τείνουν προς την εξασφάλιση δυνατοτήτων νόμιμης ε, μετανάστευσης και περιγραφής πάνω από όλα αυτής. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Ασφαλώς δεν μπορούμε να ε, υποστηρίζουμε μόνο αυτούς που μας είναι πιο αρεστοί ή πιο συμφέροντας. Πρέπει να κοιτάξουμε και τη σταθεροποίηση των περιοχών από τις οποίες έρχονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Φερρυπίν, Λιβύη, υπάρχει μια προσπάθεια για συνεργασία με τη Λιβύη. Πρέπει να ξέρετε ότι 1,5 εκατομμύρια νεκροί έχουν καταγραφεί στην ε, Σαχάρα την ίδια. Άνθρωποι που προσπάθησαν να διασχίσουν τη Σαχάρα για να φτάσουν σε ακτές της Λιβύης. 1,5 εκατομμύριο νεκροί. Τους ξεχνάμε, τους αγνοούμε. Και το μεγάλο νεκροταφείο δεν είναι η Σαχάρα, δεν είναι η Μεσόγειος, αλλά η Σαχάρα Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και όχι μόνο όταν φτάσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε πολλές ευθύνες εμείς ως ε, Ευρώπη και πολλά πράγματα να συζητήσουμε με τα κράτη προελεύσεως και τα κράτη-μέλη. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια στην Αφρικανική Ήπειρο ώστε να μπορούν να υποφεληθούν οι απλοί πολίτες. Νομίζω ότι αν μπορούμε σε κάποιε απλές αρχές όπως αυτές να συνεννοηθούμε, μπορούμε ω κοινοβούλιο να είμαστε ενωμένοι και άρα να έχουμε και μεγάλο ειδικό βάρος. Δεν μπορούμε να φροντίσουμε όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάθε γωνιά του κόσμου. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια καλή και δομημένη Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ για την Ολλανδική Προεδρία. Θέλετε να λάβετε το λόγο? Όχι. Επομένως, ας ξαναπάρει το λόγο η Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με λέτε η Επιτροπή συνέχεια, αλλά επιμένω, είμαι Ευρωπαϊκή Εξωτερική ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά είμαστε εδώ μαζί με την Επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, και είμαστε κομμάτι της Επιτροπής. Και ε, για να αναφερθώ στην τελευταία παρέμβαση, και έτσι να ξεκινήσω τη δική μου απάντηση. Είπατε ξεκάθαρα, μάλλον, δεν το είπατε έτσι σαν σκιζοφρενική κατάσταση ακριβώς, αλλά αναφέρατε ότι υπάρχουν ζητήματα συνοχής μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχουν και εντός των ε, ίδιων των κρατών μελών, μεταξύ δηλαδή Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Εξωτερικών, διαφωνίες. Γι' αυτό παρακαλώ, μελετήστε αυτή την ανακοίνωση. Δείτε τη σε ένα έγγραφο με τα θετικά και τα λιγότερο θετικά στοιχεία της, αλλά πάντως ένα έγγραφο το οποίο επισημαίνει ζητήματα που ίσως κάποια θα χρειάζονται περισσότερο να τονιστούν, κάποια ίσως λιγότερο, αλλά πάντως ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και να τα σχολιάσουν. Θα έχουν την ευκαιρία εν ώψη της απόφασης που θα ληφθεί και θα πρέπει να δοθεί και στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα μία κατεύθυνση. Παρακαλώ λοιπόν αυτή την ανακοίνωση σαν, σαν πρωταρχικό σχόλιο το λέω αυτό, μην την θείτε σαν εξαντλητική ως προς τα όσα θέλει η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Γιουνκέρ. Είναι απλώς μια απάντηση σε αίτημα του Συμβουλίου από πλευράς της Επιτροπής και της Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τίποτε περισσότερο. Αυτό γιατί κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ είναι πάρα πολύ εύλογα. Πολλά είναι πάρα πολύ εύλογα. Αλλά και εσείς κυρίες και κύριοι βουλευτές πρέπει να τα πείτε. Όχι σε μένα μόνο, αλλά και στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πρώτη μου παρέμβαση, αλλά ήθελα να κάνω το πρώτο κομμάτι της μάνας θεμελιώδους αυτής της γενικής εισαγωγικής παρατήρησης. Και τώρα περνάω στις επιμέρους ερωτήσει. Τι είναι αυτή η συμφωνία, τι σημαίνει συμφωνία, compact. αποτελεί μια διμερή, αναθεωρημένη, ένα διμερές αναθεωρημένο θεματολόγιο μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων και τρίτης χώρας, ε, με προϋποθέσεις όπως τη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της συνθήκης της Γενέβης, ε, της επαναπροώθησης και ούτω καθεξής, όπου προσδιορίζονται δηλαδή όροι που στο παρελθόν δεν ήταν τόσο σοφείς. διμερός δηλαδή. Αναθεωρούμε το πολιτικό, ε, το πολιτικό μας θεματολόγιο με την τρίτη χώρα, με θέματα και περιβάλλοντος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και δικαιοσύνης εσωτερικών. Και μετά, αυτό το διμερές θεματολόγιο πρέπει να το στηρίξουν οι συνομιλητές μας με κάθε διαθέσιμο μέσο και προχωρώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Ή την Ισία και πάλι. Και γιατί, ε, γιατί δεν είναι στο κέντρο της προσοχής. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος ότι χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Και επίσης γιατί είναι ένα κομμάτι της ανακοίνωσης με τα σχόλια για τους 360 βαθμούς κτλ. Λοιπόν, 360 μοίρες καλύτερα. Είναι κομμάτι της συμφωνίας ε, ε, είναι κομμάτι της πολιτικής γειτονίας, έχει ήδη διμερές θεματολόγιο, όπου δεσμεύεται η Τινησία σε μια σειρά από πράγματα σε αυτό ημερή διάλογο επανεξετάζουμε τα επιμέρους στοιχεία του διαλόγου. που αφορούν ε, τις ε, μεταναστευτικές ροές, τη συνθήκη της Γενέβης, τον τρόπο που θα επιλεγεί για την επαναπροώθηση, για την αντιμετώπιση της παράτυπες μετανάστευσης. Αυτά όμως είναι στόχος στράτευσης που οι ίδιοι οι Τινήσοι έχουν επιλέξει. Όρισαν δηλαδή τι μέλλον θέλουν για την Ισία για να έχουν μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη την Ισία με εθνική κυριαρχία και ως προς τη διαχείριση των συνόρων τους και χωρίς ε, παρεμβάσεις. Αυτό είναι θα έλεγα το εφιές e περισσότερα για περισσότερα, αντί για το ηλίθιο ε, περισσότερα για περισσότερα, γιατί αυτό το ηλίθιο ή ανόητο περισσότερο για περισσότερα, μόρφο μόρφο που είχαμε παλιά, ήταν να σου δίνω μερικά καρότα ή μερικά μπισκότα και να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Αυτό που λέμε όμως τώρα με την ευφυή e αυτή προσέγγιση είναι να λέμε στην Τινησία εσύ μέσα στην εσωτερική σου εθνική κυριαρχία επιλέγεις τον τρόπο με τον οποίο θα υιοθετεί τους στόχους που έχουμε ορίσει και έτσι και εγώ θα σε βοηθήσω και σε όρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου κτλ. Δηλαδή υπάρχει αιρεσιμότητα, υπάρχουν όροι, αλλά είναι αυτοδέσμευση ο ε, τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται. Εάν αποφασίσει δηλαδή την Ισία με σοβαρότητα να κάνει κάποια πράγματα που την εξυπηρετούν, που τη συμφέρουν και μέσα αυτά βάλει και τη συνιστόσα της μετανάστευσης, τότε αυτή εκουσίως ζητάει και αντίστοιχα λαμβάνει από εμά. Αυτή είναι η πτυχή, γιατί άκουσα κάποιες ε, παρεμβάσεις που αναφέρονται στην αιρεσιμότητα. Ναι, είναι πολιτική η αιρεσιμότητα. Δεν είναι η αιρεσιμότητα του τύπου αν δεν πάρεις ε, μερικούς μετανάστες ε, δεν θα σου δώσω αυτό που σου είχα υποσχεθεί ή έχω, ένα όπλο, έχω μια απειλή κρυμμένη στο μανίκι. Μιλήσατε πολύ από εσά για το ζήτημα της ε, διαφθοράς, διαφθαρμένες κυβερνήσεις, δικτατορίες και το καθεξής. Αυτό δεν μπορεί να δουλέψει φυσικά αν δεν υπάρχει δημοκρατικό καθεστώς. Πρέπει να είναι διμερείς οι σχέσεις και η αιρεσιμότητα να συμπεριλαμβάνει το γεγονός της ε, του χαρακτήρα της χώρας. Να μην έχει δηλαδή η χώρα χαρακτήρα η οποία, ο οποίος την καθιστά πηγή μετανάστευσης. Γιατί άλλο να να άμει μια πλημμύρα κτλ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις αναγκάζουν τους πολίτες τους στην φυγή. Και πολλές είναι πάμπλουτες χώρες. Πώς λέμε μην καίγεται μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Αυτό θέλω να επισημάνω για την ανακοίνωσή μας. Έχουμε στην ανακοίνωση περιλάβει την ιδέα ότι η εταιρική σχέση θα είναι 360 μοιρών, πανοραμική και ολιστική και θα μας βοηθήσει και για να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση, ε, έχοντας πρώτα να θεωρήσει την ίδια την ιδέα την αντίληψη των εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες αυτές χώρες και με αξιοποίηση των κονδυλίων για την ανάπτυξη. Και μια παρατήρηση για τα οικονομικά που ε, ελπίζω να απαντά σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Πιο πολλά χρήματα, υποσχεθήκαμε, πώς ε, θα τα διαχειριστούμε, πώς θα παρακολουθήσουμε την ε, απορρόφησή τους. Πρώτον, καταρχάς, ήδη είναι δρομολογημένα τα κονδύλια και οι μηχανισμοί παρακολούθηση από τα κράτη-μέλη, ηλεκτρικό συνέδριο κτλ. των κονδυλίων της ανάπτυξη. Αυτά ω προς την ε, παρακολούθηση. Για τα έκτακτα κονδύλια. Έκτακτα κονδύλια δεν ξέρω να υπάρχουν. Δεν έχουμε προβλέψει έκτακτα κονδύλια από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όπω σωστά υπόθηκε νωρίτερα, δεν βλέπει κανεί τα κράτη-μέλη να δίνουν υποσχέσει για όγκου οικονομικού προ την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, πίσω από την ανακοίνωση και προσπάθησα στην εισαγωγική μου παρέμβαση να το εξηγήσω, είναι και η πρόταση πως πρέπει να εξεταστεί μια νέα στρατηγική θεώρηση, ένα νέο στρατηγικό όραμα μια εξωτερική διάσταση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Και ξαναγυρνάω στο παράδειγμα της Τινεσίας. Η οποία έχει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρώπη και στην οποία σε ορισμένη χρονική στιγμή η Volkswagen σκεφτόταν να κάνει επένδυση και να αναθέσει υπεργολαβίες για κάποια ανταλλακτικά, κάποια τμήματα των αυτοκινήτων της. Ε, Ιταλός νομίζω ο Ευρωβουλευτής έθεσε ένα ερώτημα σχετικό. Να λοιπόν, η Ιταλία συγκεκριμένα έχει συμφωνία για υπεργολαβίες και franchising που δίνουν δουλειά σε 30 με 40 χιλιάδες εργαζόμενους στην Τινησία στον χώρο της κλωστή φαντουργίας. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τα αναπτυξιακά κονδύλια, δεν πολλαπλασιάζονται. 500 εκατομμύρια το αποθεματικό αναφέρεται στην ανακοίνωση, αλλά παραπάνω χρήματα δεν υπάρχουν να διαθέσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε χρήματα αρκετά ώστε να αλλάξουμε ριζικά την οικονομική διάσταση. Αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι με ένα νέο κύμα εξωτερική διάστησης επενδύσεων. φερειπήν συμφωνία ανοιχτών εθέρων με την ε, την Ισία, Ryanair, ε, German Wings ε, και άλλες low cost ευρωπαϊκές να αναπτύξουν τις πτήσεις τους, να γίνουν πολλές διωτικές επενδύσεις. Αυτό θα ήταν ένα επενδυτικό σχέδιο λοιπόν, όπως το εννοεί η ανακοίνωσή μας, προς την κατεύθυνση αυτή των ιδιωτικών επενδύσεων. Αλληλένδετα. Είναι αυτό που λέγαμε, το more for more. Εάν στο θεμερί μου πολιτικό διάλογο με την Τινησία, οι Τινήσιοι μου λένε εμεί θέλουμε την κοινωνική, οικονομική μα εξέλιξη να την ε, προσδέσουμε στην Ευρώπη, τότε ναι, θα υπάρχει και από δική μα πλευρά δέσμευση για το τι πρέπει και δεσμευόμαστε να κάνουμε. Και κάτι ακόμη ε, για την ε, νόμιμη μετανάστευση. Ποιος ανέφερε τη νόμιμη αν την ανέφερε ο Τιμ την ε, νόμιμη ω υπουργό των Εξωτερικών, ή ε, ακούσει μάλλον τον Υπουργό Εξωτερικών κάποια στιγμή και μάλιστα εγώ ήμουνα τότε εκπρόσωπο του Επιτρόπου Βιτορίνο στην, ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μιλούσαμε, όπου υπήρχε η περίφημη κοινή πρόταση ασύλου και μετανάστευση, 15 χρόνια τώρα είναι στην Τράπεζα των Συστήσεων. Τότε λοιπόν, το καιρό εκείνο, συζητήθηκε πολύ σοβαρά το πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά τρόπο ευφύη και πρακτικό την νόμιμη μετανάστευση. Άλλο οι πρόσφυγες. Εδώ δεν έχουμε νομική βάση, είναι θέματα αλληλεγγύη, ανθρωπιστικά, συνθήκη τη Γενέβη. Ωστόσο, ως προς τους παράτυπη μετανάστευση, αυτό που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι μια εξίσωση, ε, προσφορά και ζήτηση εργατικού δυναμικού. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί και να εξισορροπηθεί. Παράδειγμα λοιπόν, πριν από 15 χρόνια, την εποχή του Επιτρόπου Βιτορίνο, όπου είχε προ σταθεί μία ε, σε μια περίοδο μάλιστα κρίσης γεωργικής ε, στην Ισπανία, το Μαρόκο και άλλες περιοχές, ε, ένα σύστημα με εποχικές συμβάσεις για γεωργικές εργασίες. Παραδείγματι κάποιος από την υποσαχάρια Αφρική θα μπορούσε να πάει στην Ισπανία, την Ιταλία για τη συγκομιδή της ντομάτας και μετά να γυρνούσε πίσω. Ωστόσο κάποιες κυβερνήσεις και δι πολιτικά κόμματα την εποχή εκείνη διατύπωσαν κατηγορίες κατά της πρότασης αυτής ότι τάχα θα εκμεταλλευόταν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή θα τους φέρναμε στην Ευρώπη, θα δουλεύαν τις τέσσερις μήνες και να τους πετάγαμε πίσω. Ωστόσο η φιλοσοφία πίσω από την πρόταση ήταν να επιτρέπεται αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να δουλέψουν χωρίς να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους κατά τη διέλευση, να έχουν ασφάλιση να πληρωθούν καλά χρήματα και όχι ψίχουλα και όταν περάσουν αυτοί οι τέσσερις μήνες να είναι ευχαριστημένοι να γυρίσουν προς τις πατρίδες τους και να φροντίσουν για τις οικογένειές τους. Εδώ λοιπόν είχαμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή πρόταση, αλλά επανερχόμαστε στο πρώτο ερώτημα. Στις συμφωνίες και εταιρικέ σχέσεις με τις τρίτες χώρες δεν θέλουμε να συζητούμε μόνο επανεισδοχή ή επαναπροώθηση, έχουμε να κάνουμε με μια γενικότερη διάσταση των εξωτερικών συνόρων, μια εταιρική σχέση ότι, όπου βεβαίως ε, προβλέπεται και η επανειστοχή, ε, αλλά ταυτόχρονα και η νόμιμη μετανάστευση. Ας σταματήσω εδώ όμως. Το κύριο μου μήνυμα ήταν τα, παρακαλώ πολύ τα σχόλιά σας Βεβαίω να τα και σε μένα, βεβαίω τα δέχομαι, αλλά και προ τα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάτε ότι η ανακοίνωση προκύπτει κατόπιν εντολής του Συμβουλίου που ακολούθησε προηγούμενη εντολή, η οποία είχε και με τη σειρά της ακολουθήσει προηγούμενη εντολή και πάμε πίσω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της πρώτης έκρηξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού και θα γνωρίζετε όλοι ποια ήταν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όπου γινόταν λόγος για κάποιο είδους εισβολή και άρα θα έπρεπε να μεριμνήσουμε για τα σύνορα και τα λοιπά και τα λοιπά και να αναπτύσσουμε μια εξωτερική διάσταση. Όχι να τους γυρίσουμε πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η πολιτική αντίδραση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και γι' αυτό σας καλώ να ρίξετε μια ματιά και πάλι στα ε, συμπεράσματα των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Οκτωβρίου του 2015. 15 αν δεν απατώμε, Οκτωβρίου. Και διαβάστε τα συμπεράσματα που είναι τα συμπεράσματα των κρατών μελών. Και αυτό είναι το μήνυμα που αποστέλουν σε εμά τα θεσμικά όργανα. Αυτή είναι η εντολή που μα έδωσαν. Εκεί θα δείτε το περίφημο more for more ή less for less, με την έννοια του εάν δεν συνεργάζεται για την επανεισδοχή, τότε ε, έχετε συνέπειες. Εδώ τώρα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, εταιρική σχέση, υπευθυνότητα και συνεργασία και από την άλλη πλευρά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της επανεισδοχής, αλλά, γιατί απαιτείται, αλλά είναι πολύ ευρύτερα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ανακόνηση. Ευχαριστούμε κύριε Γκαμπρίτσε. κύριος από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Να συμπλώσω τα τεχνικά θέματα. Ε, τα γενικά ε, θέματα τα, τα παρουσίασε πάρα πολύ ο Λιονέλο. Καταρχάς, το θέμα της εταιρική ε, σχέσης του συμφώνου. Ποια είναι η προσέγγισή μας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αναθέσουμε σε τρίτους τις δικές μας ευθύνες για τα σύνορά μας. Αυτό που θέλουμε και κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το δυναμικό των χωρών αυτών να προστατεύουν τα δικά τους σύνορα. Και οποτεδήποτε πάτε σε αυτές τις χώρες θα ακούσετε να λένε ότι θέλουν κάτι τέτοιο. Γιατί καμία χώρα στον κόσμο δεν θέλει οι λαθρέμποροι, οι διακινητές να περνάνε τα σύνορά της χωρίς έλεγχο. Γιατί οι διακινητές ε, δεν διακινούν μόνο ανθρώπους, αλλά οποιαδήποτε αγαθά. Επίση, θέλουμε να αναλάβουμε προφανώς τις ευθύνες μας για τη διεθνή προστασία. Κανένα δεν προτείνει να σταματήσουμε να το κάνουμε και να μην λαμβάνουμε ε, πραγμα... και να μην προστατεύουμε πραγματικούς πρόσφυγες, γνήσιους πρόσφυγες. Αυτό που προτείνουμε είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες νομικές και νόμιμες οδούς ε, στα πλαίσια του συμφώνου, συν εγκατάσταση ε, ή επανεγκατάσταση. Δεν αποφεύγουμε τις ευθύνες μας λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως φεύγουν από πολέμους, αλλά ακόμα και αυτοί προτιμούν να παραμένουν κοντά στις χώρες προέκλευσή τους, όπως παραδείγματος χάρη η Αιθιοπία και Λίβανο. Είναι σημαντικό να να εγκατασταθούν εκεί που επιλέγουν. Γιατί αν δεν υπάρχουν συνθήκε για να εγκατασταθούν, θα πρέπει να φύγουν πιο μακριά από την χώρα προέλευσή του. Δεν είναι ότι του εμποδίζουμε να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκε ε, για να παραμείνουν εκεί που επιλέγουν να παραμείνουν. Για τις εξελίξεις ε, δεν νομίζω ότι εμεί από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μπορούμε να σχολιάσουμε τα εργαλεία κτλ. Ας δούμε όμως τις ευκαιρίες. Φυσικά θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να συνεργαστούμε και να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας στα πλαίσια μια εταιρική σχέση, να δούμε τι είναι απαραίτητο να γίνει και τι δεν είναι. Δεν ψάχνουμε να κάνουμε μόνο περικοπές και να τιμωρήσουμε ας πούμε. Όχι, θέλουμε να ακούσουμε και να καταγράψουμε και να δώσουμε αυτό που θέλουν αυτές οι χώρες. Τώρα, αν θα πρέπει να είναι τεχνική αρρωγή αυτή ανταλλαγή των πρακτικών κτλ. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση δυναμικού. Είμαστε και από τη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων, προσωπούμεθα δηλαδή εκεί, και από άλλες γενικές διευθύνσεις, ε, για να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των τρίτων χωρών. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τις παρεμβάσεις τους. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σα διάταξης, αλλά πρωτού συμβεί αυτό, να ανακοινώσω ότι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διαταξή για σήμερα το πρωί το σημείο 15 θα αναβληθεί διότι έχει καθυστέρηση η υπεύθυνη του σημείου αυτό η κυρία Φαγιών ίσως να το δούμε αύριο το πρωί και τώρα να περάσουμε στο θέμα του πώς έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ψηφίσαμε στις 30 Μαΐου την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μας και έκτοτε έχουν αρχίσει τριμερείς διάλογοι. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην, στον εισηγητή, στον κύριο Πάμπριξ, για να μας ενημερώσει για το πώς έχουν προχωρήσει οι τριμερείς διάλογοι. Σε ευχαριστώ Κίνγκα. Μεγάλο μέρος της δουλειάς έχει γίνει σε ό,τι αφορά τι συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή, την Ακτοφυλακή και την σχετική πρόταση. Να θυμίσω στους συναδέλφους, για όσους δεν παρακολουθούν καθημερινά τα θέματα αυτά ίσως, ότι πρόκειται για ένα άκρος σοβαρό από στρατηγικής, πολιτικής και θεσμικής σκοπιά ζήτημα για όλους μας. Σκοπό έχει να ενισχύσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της Frontex και να εξεύρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη φάση η Ευρώπη ε, γνωρίζει άνευ προηγουμένου μεταναστευτικές πιέσεις, μια κρίση που πρωτόγνωρη και επίσης ε, απειλές ε, εγκληματικών ενεργειών, τρομοκρατικών ενεργειών λόγω της αστάθειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Από αυτήν την οπτική γωνία δεν έχουμε και πολλές ε, δυνατότητες, ούτε περιθώριο ελιγμών σε σχέση με τα εξωτερικά μας σύνορα και τη διαχείρισή τους. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα εντός αυτού του περίπλοκου θέματος που πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Εάν τα δείτε και από την οπτική γωνιά των ε, χωρών μελών και των Ευρωπαίων πολιτών, που εκπροσωπεί ακριβώς το Κοινοβούλιο, όλοι περιμένουν από εμά να καταλήξουμε εδώ σε μια απόφαση η οποία να μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και θα πρέπει κι εμείς ως θεσμικό όργανο, ως Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς αυτό να αποδείξουμε, ότι μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση που θα επηρεάσει θετικά τα δικαιώματά μας, την ασφάλεια των πολιτών και θα ε, εγγυηθεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, της προδιαγραφής για όλους αυτούς τους καψερούς που προσπαθούν να φτάσουν ε, στις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να είναι ασφαλείς και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το πώς έχουν προχωρήσει τριμερείς διάλογοι, να σας ενημερώσω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να έχουμε πέντε συναντήσεις τεχνικού περιεχομένου και τρεις τριμερείς διαλόγους. Ο τελευταίος ολοκληρώθηκε χθε. Να πω ότι πετύχαμε σημαντική πρόοδο και πραγματικά χάρη στην σκληρή δουλειά των συνεργατών και βοηθών μας και βεβαίως με την πλήρη συνεργασία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών μας. Απλώς δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους και για την ε, δουλειά τους και για την προσέλευσή τους. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταλήγουμε σε συμφωνία, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να αποβάλουμε ένα καλό έγγραφο ε, και να γιορτάσουμε την νίκη μας και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι προσεγγίζουμε μια ε, συμφωνία με το Συμβούλιο για πολλά σημεία και πολύ σύντομα να τα απαριθμίσω και να τα εξηγήσω γιατί είναι τα θετικά. Το πρώτο είναι το άρθρο 4, η έννοια της ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε συμφωνήσει εδώ. Επίσης, σε γενικές γραμμές έχει συμφωνηθεί και γίνει ε, αποδεκτό ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η λογοδοσία είναι κάτι που πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό θα αυξήσει και την αξιοπιστία του θεσμικού μας οργάνου και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από την πλευρά των δικαιωμάτων. Να πούμε κάθε ειλικρίνεια ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή Είχαν αμφιβολίε για πολλά ζητήματα, για μια σειρά από ζητήματα εδώ, αλλά καταφέραμε να περάσουμε τη δική μα άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, παρουσία των λεγόμενων ε, αποσπασμένων αξιωματικών, το άρθρο 11, ε, εδώ μπορέσαμε να προχωρήσουμε παρά τους ενδιασμούς του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Καταφέραμε να τους εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και να εργάζονται σε τρίτες χώρες, διότι πραγματικά θα διευκολύνουν τη συνεργασία μας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούμε καταστάσεις όπου αποτελεσματικά μπορούμε να διαχειριστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα στο μέλλον και εγκαίρως να παράσχουμε ε, έκτακτη βοήθεια, εάν δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Οπότε αυτοί οι αξιωματικοί σύνδεσμοι που ήταν η δική μας η πρόταση ακριβώς για αυτόν τον τριμερή διάλογο είναι σημαντική και η παρουσία τους επίσης για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και σε σχέση με, το, μετριακή δημόσιο που μας υπερβαλεί η Επιτροπή. Το νέο θέμα στο οποίο μπορώ να, σημειώ, να πω ότι σημειώσω με πρόοδο είναι η έκθεση ε, του κατά πόσον είναι ευάλωτες κάποιες χώρες. Δηλαδή, οι εξωματικοί σύνδεσμοι θα κάνουν τέτοιε εξελογήσει στο επίπεδο των συνόρων και θα υπάρχει συμπληρωματικό μηχανισμό ε, που θα σχετίζεται απευθεία με το σύστημα Schengen. Δηλαδή, θα υπάρχει παραλληλισμό και συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι και πάλι θα έχουμε καλύτερη κατανόηση και έγκαιρη γνώση για το τι συμβαίνει αλλού. Επίσης προσπαθούμε να επιτύχουμε πρόοδο στα θέματα του τεχνικού εξοπλισμού διότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για να δοθεί έγκαιρη βοήθεια και ανθρώπινη πόρη ε, στην συνοφυλακή και ακτοφυλακή, αυτό θα είναι μισή επιτυχία. Ε, Πολλέ φορέ, όταν οι άνθρωποι αυτοί πάνε να εργαστούν σε μια τρίτη χώρα και δεν έχουν τα τεχνικά μέσα, δεν μπορούν να φέρουν ει πέρα στο καθήκον του. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει παράλληλη στήριξη από του ανθρώπινου πόρους και η ακατάλληλη τεχνική υποστήριξη. Προφανώς εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ως προς το ποιες χώρες θα παρέχουν τα τεχνικά ε, μέσα. Αφήσαμε χρόνο στο Συμβούλιο για να δει πώς θα το καταφέρει αυτό, αλλά Ελπίζω ότι θα βρει το Συμβούλιο εγκαίρως να βρει τρόπο για να απαντήσει και στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό της έγκαιρης έκτακτης βοήθειας. Όσο για τους 150.000 εξηματικούς μάλλον 1.500, για τους 1.500 συνεργοφύλακες και ε, εργαζόμενους στην ακτοφυλακή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει ο... η συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δεν καταλαβαίνουμε εδώ και τη συλλογιστική της επιχειρηματολογίας του Συμβουλίου. Ε, ε, σε στιγμή ανάγκης θα μας βοηθήσει να μπορούμε να ζητούμε έναν υψηλό αριθμό έκτακτων αποσπασμένων εφόσον χρειαστεί διότι δεν μπορούμε να παγώσουμε το ανώτατο αυτό όριο στα 1500 άτομα αναγκαστικά. Ποιο τι θα συμβεί στο μέλλον. Μιλάμε για έναν οργανισμό που δημιουργούμε σήμερα με τι σημερινέ συνθήκε, αλλά θα πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη συνδρομή και βοήθεια στα θέματα αυτά για την ερχόμενη δεκαετία τουλάχιστον. Επίση, ε, επιτύχαμε ε, θεμελι... ουσιαστική πρόοδο στα θεμελιδία δικαιώματα. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Υπάρχει μνήα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο άρθρο 1 στην ε, ουσία δηλαδή, στο ίδιο το περιεχόμενο και το πεδίο του κανονισμού που είναι κάτι σαν ομπρέλα για ολόκληρο τον κανονισμό. Επίσης ε, για τους πόρους που χρειάζονται για τα ανθρωπιστικά ζητήματα και εκεί υπάρχει μια η ανάγκη πόρων η ανάγκη ανθρωπιστικής στήριξης είναι κάτι που κάθε πολιτική δύναμη εδώ, εντός ή εκτός των τείχων του Κοινοβουλίου, είναι κάτι που νομίζω θα το αναγνωρίσει, ότι δεν έχουμε δώσει μικρή σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι μας ανησυχούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό και εν τέλει έχουμε στηρίξει και την ε, ε, δημιουργία, την ίδρυση αυτού του οργανισμού. Βεβαίως δεν υπάρχουν δρόμοι χωρίς ε, κάποιες ανομαλίες. Υπάρχουν ακόμη κάποιες δυσκολίες, οι τριμερείς διάλογοι θα συνεχίσουν, το ίδιο και οι ε, τεχνικές συζητήσει. Κάποια από τα τεχνικά ζητήματα στα οποία έχουμε σκοντάψει είναι το εξής. Προβληματικό ανεπίλητο ακόμη ζήτημα της κατεπίκουσας δράσεις βάσει του άρθρου 18. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να στηρίξει το Συμβούλιο ώστε να λαμβάνει εκείνο αποφάσεις, αλλά αυτό μας ζητήθηκε. Δεν συμφωνώ με το Συμβούλιο. Τι θα συμβεί εάν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να συνεργαστεί. Είναι βέβαια υποθετικό το σενάριο, γιατί υπάρχει και κοινή λογική ε, της ε, κάθε χώρας μέλους, την οποία επαφιόμαστε, και Επίσης ελπίζουμε ότι οι χώρες θα ζητούν με εύλογο τρόπο βοήθεια. Αλλά το Συμβουλίο θεωρεί ότι σε τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να επιτρέπεται ο εσωτερικός έλεγχος συνόρων. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση. Εδώ ακόμη δεν έχουμε συμφωνία. Να πω όμως ότι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή θυμίζουν ότι δεν μπορούμε να πεινοήσουμε ένα θηρίο, μια τίγρη και να τη στείλουμε κατευθείαν και στον φοντίατρο να τη βγάλουμε όλα τα φόντια. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομοθέτες, εφόσον χαράζουμε νομοθεσία, πρέπει να φροντίζουμε η νομοθεσία που χαράζουμε να ακολουθείται όλος, να γίνεται σεβαστή. Ιδάλλως δεν έχει νόημα. Αυτή είναι η δική μου ισχυρή πεποίθηση. Πιστεύω ότι η κοινή λογική πρέπει να πρετανεύσει. Το Συμβούλιο θα ήθελε να αφαιρεθεί το coast από τον τίτλο. Διότι ακόμη και αν δεν είναι νήσος η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, νερά και μάλιστα ταραγμένα και τρικυμισμένα έχουμε πολλά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να το αφήσουμε αυτό στον ε, τίτλο. Θα βρούμε ίσως μια λύση για να λύσουμε το θέμα αυτό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο δεν έχουμε πετύχει συμφωνία είναι ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή για θεσμικά, και τα θεσμικά ζητήματα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα σημείο εξισορρόπηση μεταξύ των εξουσιών του εκτελεστικού διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου που θα εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Ακόμη εξετάζουμε ενδεχόμενες συμβαστικές λύσεις εδώ, αλλά είναι σαφές ότι ό,τι και αν γίνει, όπως και αν καταλήξει αυτή η συζήτηση, ο, ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα έχει ενισχυθεί εν τέλει. Και είναι και αυτό σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι τα δικαιώματα είναι και δική μας ευθύνη. Και άλλο ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε συμφωνία είναι το τμήμα για τις επιστροφές. Ο οργανισμός θα έχει αυξημένε αρμοδιότητες ό,τι αφορά τις επιστροφές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή. δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μία άποψη κοινή. Οι επιστροφές είναι ζωτικό και αναπόσπαστο τμήμα του εγγρόφου. Δεν μπορεί να μην έχουμε μια φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη ε, κάλυψη του θέματος των επιστροφών στο κείμενο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας, τους ε, βοηθούς μας, όλο μας το τεχνικό προσωπικό και τους διερμηνείς μας που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούμε, μπορούν για να πετύχουμε μια συμφωνία επί Ολλανδικής ε, Προεδρίας. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε, αλλά διασφαλίνοντας τα σημαντικότερα σημεία για το Κοινοβούλιο και βεβαιωνόμενοι ότι θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του οργανισμού αυτού και ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλο του μήνα θα είμαι σε θέση να σα ενημερώσω ξανά για επίτευξη συμφωνία. Και ελπίζω ότι θα συμπεριλάβουμε αρκετά από τα επιτεύγματά μα για τα θεσμικά μα όργανα και όλο ιδιαίτερω για το Ευρωκοινοβούλιο μεταξύ των επιτυχιών μα. Το πλέον σημαντικό. Ο κανονισμός που προβλέπει ένα αποτελεσματικό και δραστικό οργανισμό για να μπορεί να συνδράμει τις χώρες μέλη είναι ο στόχος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να επιληθεί το ζήτημα. Να μην φανταστούμε ότι αυτό θα αποτελέσει πανάκια, αλλά εάν δεν μπορούμε να χειριστούμε ένα τέτοιο ζήτημα, ε, το ερώτημα παραπαίνει τι μπορούμε τελικά να κάνουμε στην ώρα του και πότε επιτέλους θα το κάνουμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, μην το ξεχνάμε και είναι και σημαντική και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις ή να ακούσω σχόλια ή ευχές για την καλή συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάμπριξ για τη δουλειά σας. Θα δώσω λόγο στους κοιόδης ηγητές. Λίδιν Μιούλερ θέλετε να πάρει το λόγο. Ναι. Σύντομα. Συμφωνώ με την ε, έκθεση του εισηγητή. Ε, δουλέψαμε και εντατικά και σε αγαστή συνεργασία. Έχουμε ε, ένα ή δύο-τρία εμπασπιπτώσει κρίσιμα σημεία που χρειαζόμαστε να συμφωνήσουμε προκειμένου να συμφωνήσουμε τελικά. Από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε καλούς συμβασμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Χάρη στον εισηγητή που δούλεψε πολύ έντονα γι' αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το βασικό πρόβλημα κατά την απόψή μας είναι το θέμα της, των επιστροφών και όλων των επιχειρήσεων επιστροφών. Και ο ρόλος της συνοριαφυλακής σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να εμφαν... Ε, τονιστεί. Η συνοριοφυλακή δεν μπορεί να γίνει πραγματικός οργανισμός ή φορέας επιστροφών. Έτσι. Φυσικά, ε, οι επιστροφές είναι σημαντικό τμήμα της διαχείρισης των συνόρων, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Είναι ένας τομέας από το οποίο ε, εργαζόμαστε ακόμα για να πετύχουμε συμβιβασμό και είμαι πολύ, πολύ σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα φτάσουμε σε αυτό το συμβασμό. Ευχαριστώ κύριε Νίτερ Κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αντικαταστήσω την Νάταλη Γκρισπέκ που δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ και θα προσπαθήσω να μιλήσω γαλλικά για πρώτη φορά στην Επιτροπή. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του δούλεψε εργοδός. Α, ήρθε και η Ναταλή. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων η Ναταλή μια στιγμή να πάρει λίγο μια ανάσα. Θέλει να τονίσει διάφορα σημεία λοιπόν η Ναταλή. Καταρχάς, να κάνουμε ε, προσπάθειες ε, έρευνας και διάσωσες σε... και αυτές οι αποστολές να είναι τμήμα των καθηκόνων της νέας, του νέου οργανισμού της Frontex για την δομή του οργανισμού αυτού. Ε, το Κοινοβούλιο και κυρίως η ομάδα φιλελεύθερων υποστηρίζει από την αρχή τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, ε, ισχυρής ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Θα έχει σημαντικές εξουσίες η διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό θα πρέπει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να έχουν πραγματικό λόγο σε, αυτή, σε αυτόν τον διορισμό. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Αταλή να τα πει με, της, με τα δικά της λόγια. Ε, καλημέρα σε όλους. Καταρχάς να ευχαριστώ πάρα, να ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σεσίλια, η οποία μίλησε την διπλωματική γλώσσα του Μολιέρου με το ταλέντο που όλοι ξέρετε ότι έχει και που τελευταία στιγμή δέχτηκε να παρουσιάσει α, λίγα στοιχεία σε αυτή τη γρήγορη συζήτηση που έχουμε. Ε, συγγνώμη, αλλά ε, αντί για δυόμιση ώρες ε, συνάντησα ένα α, αγριογούρουνο ε, συμφόρηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση ε, είχα πολλά εμπόδια και τελικά για δυόμιση ώρες έκανα τέσσερις. Σας ευχαριστώ λοιπόν που δεχτήκατε να την, τη Σεσίλια δηλαδή που ήθελα να με αντικαταστήσει. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους και εισηγητές, κυρίως για την αποφασιστικότητα και ισχυρή βούλησή τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική και επί της ουσίας, αλλά και είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση γιατί ε, ενώ οι πολίτες συχνά δεν ξέρουν τι κάνει η Ευρώπη, αυτή την έκθεση την παρακολουθούν. Προσπαθούν να καταλάβουν και περιμένουν και απαντήσεις. Η Σεσίλια το είπε. Οι απαντήσεις μέσω αυτού του φακέλου θα είναι καθολικές. Δεν θα επιτρέψουν όμως με αυτή την αναθεώρηση να λυθούν όλες οι προκλήσεις, κυρίως οι μεταναστευτικές ε, προκλήσεις, γιατί αυτό δεν είναι το μόνο μέσο. Ε, ευχαριστώ τον Άρτης ε, για τη δουλειά που έκανε, κατα, καταπληκτική δουλειά. Και η Σεσίλια μίλησε για τα δύο σημεία, και την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, που για τους περισσότερους σκιώδεις ηγητές θα πρέπει να μπει ε, στις αποστολές αυτού του νέου οργανισμού, αυτής της νέας υπηρεσίας και φυσικά το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα το συζητήσουν. Ε, Επίση, ευρωπαϊκό χαρακτήρα, το είπε η Σεσίλια. Και τρίτο σημείο, πολύ γρήγορα τα λέω όλα αυτά, είναι όλα αυτά που αφορούν τις επιστροφές Δηλαδή τι διατάξει για τις επιστροφές Οι φιλελεύθεροι θέλουν μια, ε, μια πολιτική επιστροφών αποτελεσματική και κυρίως και αυτό το λέμε σε κάθε συνεδρίαση και τεχνική και πολιτική του Τριλόγου, να συνοδεύεται από όλε τι ευρωπαϊκέ εγγύησει μη επαναπροώθηση και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια όμως του νέου ρόλου της Frontex σε ό,τι αφορά τις ε, επιστροφές, το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός βοηθάει τα κρατημέλη στις επιχειρήσεις ε, επιστροφών είναι κάτι πολύ σημαντικό και καινούριο και στα πλαίσια των συζητήσεων για την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής το να δοθεί δηλαδή αρμοδιότητα στη Frontex ώστε να βοηθήσει τις επιστροφές από τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα, αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην πάμε να ασχοληθούμε τώρα άλλα. Ε, να σεβαστούμε τα δικά μας κριτήρια για να μην χάσουμε την αποτελεσματικότητά μας και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις ε, επιστροφών που θα διεξάγονται από τρίτη χώρα σε τρίτη χώρα. Ελπίζω να τα είπα ξεκάθαρα. Ε, μακρηγόρησα λιγάκι, συγγνώμη, ε, φταίνουν και οι περιστάσεις. Ε, σας ευχαριστώ που δώσετε περισσότερο χρόνο στην ομάδα μου. Ευχαριστώ Ναταλή και ευχαριστώ τη Σεσίλια. Μπράβο Σεσίλια. κυρία Μπιόρκ. Ναι, ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Όπως ξέρετε, ο Λιγκού έχει σοβαρές επιφυλάξεις όλη αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής. Πρέπει να διαγραφεί κάθε αναφορά σε ακτοφυλακή επίσης. Ο σκιώδης ηγητής Αλμπιόλ πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσει το ζήτημα των επαναπροωθήσεων. Εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε καταψηφίσει αυτή την ε, ιδέα να αναλάβει αυτή, μια, αυτή η super ε, Frontex την ε, επαναπροώθηση από τη μία τρίτη χώρα στην άλλη, από την Τουρκία προς το Ιράκ, παραδείγματι. Ε, το έχει και αποφασίσει το Κοινοβούλιο αυτό και πρέπει αυτή ε, τη θέση να την στηρίξουμε. Έχει καταψηφίσει αυτή την πρόταση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να θεσπιστεί μια αρχή η οποία θα έχει να επιβάλλει επαναπροώθηση μεταξύ τρίτων χωρών. Γιατί τότε δεν θα γίνεται σεβαστό το δίκαιο του ασύλου. Ευχαριστώ. Επιτροπή. Θέλετε το λόγο, όχι. Πάμπριξ, όχι. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλές διαπραγματεύσεις, καλά αποτελέσματα. Μας περισσεύουν 10 λεπτά μέχρι την ώρα των ψηφοφοριών. Διάλειμμα λοιπόν. Και ξαναρχίζουμε στις 11.30. ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση ε, ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust. Uh, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Για να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Εύκολες είναι. Δύο μόνο. Μία ερώτηση προς την Επιτροπή και μία προς το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust. Εάν μπορείτε όλοι καθίστε. Και θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή για την θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και την Eurojust. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Προφανώς εγκρίνεται. Και ερώτηση προ το Συμβούλιο για το ίδιο θέμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτά εγκρίναμε τις διερωτήσεις. Αυτά για σήμερα το πρωί. Θα έχουμε πολύ πιο δύσκολες ψηφοφορίες την επόμενη εβδομάδα, τρίτη πρωί. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Όπως ε, σας είχα πει, ε, θα κλείσουμε την ε, σημερινή μας συνεδρία στο πρωί στις 12. Η έκθεση της κυρίας Φαγιών αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Τελευταίο σημείο για την πρωινή μερίσια διάταξη. Κυρία Μακοβέη, με συγχωρείτε μπορείτε να τα ξαναπείτε, γιατί έχει θόρυβο στην αίθουσα. Η έκθεση φαγιών για το 25 αναβλήθηκε. Ναι, γιατί η, το αεροπλάνο της κυρίας Φαγιών είχε καθυστέρηση, οπότε δεν είναι θα έρθει και ζήτησε να ε, προγραμματιστεί εκ νέου. Μάλλον δεν προλαβαίνουμε με το χρονοδιάγραμμα αύριο, οπότε θα πάει την επόμενη εβδομάδα. Η γραμματεία πάντως το ε, εξετάζει. Θα ολοκληρώσουμε την πρωινή συνεδρίαση στις 12. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Να συνεχίσουμε λοιπόν την πρωινή μας συνεδρίαση με την παρουσίαση της τελευταίας εκδοχής του τελικού σχεδίου μελέτης της ομάδας Μιλιού οι οποίοι μελέτησαν το θέμα που ζήτησε η Επιτροπή μας. Εκτίμηση αντικτύπου εισοδιωτών τροποποιήσεων που διεξήθη την κατανάθεση τη μονάδα εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου τη Υπηρεσία Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Για το δικαίωμα δικαστική συνδρομή για υπόπτου, ή κατηγορουμένου σε ποινικέ διαδικασίε και σε διαδικασίε εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, μαζί με μια συνολική μελέτη αντικτύπου. Να ακούσουμε τώρα τα πορίσματα της μελέτης αυτής αντικτύπου και ο λόγος σε πρώτη φάση στην κυρία και μετά η κυρία Νταλαπότσα από την ομάδα Μιλιέ. Πρώτη, η κυρία Μαριακή Γκρίβα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να υποβάλω αυτή τη μελέτη αντικτύπου των τροποποιήσεων ε, κατόπιν της, ε, ε, του αιτήματο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ πολύ γρήγορα το πόρισμα αυτή τη Επιτροπής. Η υπηρεσία εξάντε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αιτήματος τη Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διεξήγα για την έκθεση αυτή. Για τι δικέ μας ουσιώδει τροποποιήσει και για το κατά πόσο είναι απαραίτητε για την νομική διαδικασία. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μα ζήτησε να εξετάσουμε τον αντίκτυπο 7 ουσιώδων τροποποιήσεων που συμπεριλαμβάνονταν στην έκθεση ε, του κυρίου ε, Αγιών από, την, από το Μάιο του 2015. 29, 31, 34, 33 και 35. Όπως προκύπτει από το εγχειρίδιο για τις μελέτες αντικτύπου του Ευρωκοινοβουλίου, ε, οι τροποποιήσεις αυτές βασίστηκαν στα όσα όρισε η Επιτροπή Λίμπη. Λίμπε. χρησιμοποιήθηκαν αυτά που συμπεριλάμβανε και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποίησαμε τις υπηρεσίες της ομάδας Μιλιέ, η οποία βασίζεται στην, ε, ε, στις Βρυξέλλες και έχει μακρά σχέση συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η έκθεση φτάνει στα τελικά της στάδια σύντομα και θα διατεθεί στην Επιτροπή σας. Τα βασικά πορίσματα θα, συμπε... θα παρουσιαστούν σήμερα από την κυρία Βερτζίνια Νταλαπότσα, νομική σύμβουλο του Μιλιέ, και την κυρία Ανιέσκα Μαρκόφσκα, σύμβουλο επιθεματών πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαγιάκη. Ξεκινάμε την παρουσίαση των στόχων της μελέτης αυτής. Η μελέτη σκοπό έχει να αποτιμήσει τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο των των τροπολογιών, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των τροπολογιών στα θεμελιώδη δικαιώματα, των υπόπτων και κατηγορουμένων και να αναλύσει εναλλακτικά σενάρια για τις τροπολογίες 31 και 42 με σκοπό να αντικατοπτρίσει τι διαφορετικέ θέσει των τριών θεσμικών οργάνων, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπή και του Συμβουλίου. Η μελέτη βασίστηκε στην μελέτη, την έρευνα της βιβλιογραφία και στι συζητήσει με του ενδιαφερομένου. Έγινε μία μελέτη και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες για θέματα νομική, νομικού περιεχομένου. Κάναμε ανάλυση ποσοτική η οποία βασίστηκε στα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου της Επιτροπής και καλύπτει τα 28 κράτη-μέλη και ταυτόχρονα ποιοτική ανάλυση η οποία στηρίχθηκε σε 10 κράτη-μέλη. Λόγω της έλλειψης δεδομένων και του σύντομου χρονοδιαγράμματος του όλου προγράμματος η ποσοτική μας ανάλυση έγινε μόνο για τις τροπολογίες 41 και 44. Ένα από τα βασικά ζητήματα της νομικής, της δικαστικής συνδρομής είναι το γεγονός ότι τα εθνικά πρότυπα και οι προδιαγραφές διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό οδηγεί σε ελλείμματα ως προς την παροχή δικαστικής συνδρομής. Βάσει της ανάλυσής μας, η έγκριση αυτών των τροπολογιών θα έχει θετικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των ε, κατηγορουμένων και υπόπτων. Οι τροπολογίες θεωρούν την δικαστική συνδρομή ως ζωτικό στοιχείο ενός δίκαιου δικαστικού συστήματος και θέλουν και στην πράξη να παρέχεται το δικαίωμα σε πρόσβαση σε συνήγορο από τους ε, Ευρωπαίους. Ε, βέβαια, επιφέρουν και κάποιο κόστος οι τροπολογίε αυτές, όμως θα υπάρχει και μια σειρά από ωφέλη. Ένα εύρυθμο δικαστικό σύστημα επιτρέπει σε ευθυγράμμιση των διαδικασιών, μειώνει το χρόνο που περνούν οι κατηγορούμενοι σε κέντρα κράτηση και περιορίζει τον αριθμό άδικων καταδικών, καθώ και μειώνει τον υπερπληθισμό των σοπονιστικών ιδρυμάτων και την συμφόρηση στα δικαστήρια. Κάποια από τα ωφέλη είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν σε νομισματικούς όρους και εδώ μιλώ κυρίως για το ωφέλιμα της αποφυγής άδικης κράτησης ή των άδικων καταδικών. Ακόμη όμως και αν τα δούμε σε νομισματικούς όρους και είναι δύσκολο να τα μετρήσουμε, ε, αυτό δεν ε, σημαίνει ότι δεν πρέπει να εγκριθούν οι τροπολογίες τα βασικά πορίσματα της μελέτης. Τροπολογία 29. σκοπός είναι να διευρυνθεί το πεδίο της οδηγίας σε κατηγορούμενους και υπόπτους, ώστε να μην τους στερείται η ελευθερία και να τους παράσχεται τακτική δικαστική συνδρομή σε αντίθεση με την προσωρινή. Ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτή τη τροπολογία. Διευρύνοντα την δικαστική συνδρομή σε άτομα που δεν του στερείται η ελευθερία, αλλά που μπορεί να είναι αντικείμενο ανάκριση, να συμμετέχουν σε κάποια ανακριτική διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι προστατεύονται περισσότερο τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Θα εκπροσωπούνται νομικώ και υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους σε μια δίκαιη δίκη. Η διάταξη της τακτική δικαστική συνδρομή, πέραν της προσωρινή, διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε συνήγορο και το δικαίωμα σε δίκαιη εκδίκαση καθ' όλη τη διάρκεια τη δίκη. Άρα πριν και μετά την απόφαση υπάρχει μια, ένας έλεγχος αιρεσιμότητας. Η τροπολογία 29 ε, επιτρέπει καλύτερη ευθυγράμμιση των ε, εξορθολογισμών των διαδικασιών με ελάχιστα πρότυπα για την τακτική δικαστική συνδρομή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει εξοικονόμηση από τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών. Ταυτόχρονα είναι η πλέον δαπανερή τροπολογία. Βάσει τη εξέτασή μα, το κόστο εκτιμάται στην ψαλίδα 244 έως 386 εκατομμύρια ευρώ ετησίω ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός αυτός καλύπτει 61 εκατομμύρια λόγω της διεύρυνσης του πεδίου σε άτομα που δεν τους στερείται η ελευθερία τους και κατά προσέγγιση 180 εκατομμύρια λόγω της διεύρυνσης του πεδίου στην τακτική δικαστική συνδρομή. Τροπολογία 31. Εδώ αποκλείονται τα ίσονα σημασία αδικήματα από, την, από το πεδίο τη οδηγία σε δύο περιπτώσεις. Όπου μία κύρωση μπορεί να επιβληθεί από αρχή, άλλη από ποινικό δικαστήριο. Και δεύτερον, όταν η στέρηση τη ελευθερία δεν μπορεί να επιβληθεί ως κύρωση. Η δικαστική συνδρομή θα παράσχεται σε όλε τι δίκε μπροστά και ενώπιον ε, ποινικού δικαστηρίου. Ποιο ήταν αντίκτυπο αυτών των τροπολογιών. Τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων θα προστατεύονται καλύτερα σε αυτά τα κράτη-μέλη, όπου η δικαστική συνδρομή αποκλείεται για τα ίσονα σημασία αδικήματα. σε άλλα κράτη όπου δεν υπάρχει αποκλεισμό από την δικαστική ε, συνδρομή σε περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αδικήματος, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ή μπορεί να περιοριστεί η δικαστική συνδρομή για κάποια ίσονα σημασία αδικήματα, ιδίω για αυτά που χειρίζονται αρχέ άλλε από τα ποινικά δικαστήρια. Αυτό ο ενδεχόμενο περιορισμό τη δικαστική συνδρομή για ίσονο σημασία αδικήματα θα φέρει εξοικονόμηση σε επίπεδο 0,2-11% του κόστου τη συνολική δικαστική συνδρομή για άτομα που δεν του στερείται η ελευθερία του. Τροπολογία 39. Περιορισμός τη δυνατότητα των κρατών μελών να ε, ζητήσουν αποζημίωση για το κόστο ε, δικαστική συνδρομή. ή ο περιορισμός αυτός θα βασίζεται σε δύο προϋποθέσεις. Πρώτο, η τελική απόφαση που καθορίζει ότι κάποιος δεν πληρεί τα κριτήρια ρεσιμότητας για την τακτική δικαστική συνδρομή είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ψευδείς πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου ή υπόπτου. Στι δύο αυτέ περιπτώσει τα κράτη-μέλη μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα παροχή δικαστική συνδρομή και να πάρουν πίσω το κόστο αυτή. Αυτή η τροπολογία μάλλον θα μας φέρει σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που θα παίρνουν δικαστική συνδρομή, διότι θα μειωθεί ο κίνδυνος να του ζητηθεί πίσω το κόστος. Το κόστος αυτής της επιλογής για τα κράτη-μέλη έχει εκτιμηθεί σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 15% του κόστους που ανακτούν αυτή τη στιγμή. Ανάλογα με τους όρους και τις προποθέσεις που πληρούνται. Τροπολογία 41. Ανεξάρτητη αρχή μια απόφαση να παράσχεται δικαστική συνδρομή και να διοριστεί συνήγορος θα λαμβάνεται από ανεξάρτητη αρχή. Η τροπολογία αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στο δικαίωμα πρόσβασης συνήγορο, σε δίκαιη εκδίκαση, στην ε, ισοδικία και την πρόσβαση σε συνήγορο καθώς και το τεκμήριο ε, θα πρέπει ε, η ανεξάρτητη αρχή να αποφασίσει το διορισμό συνηγόρου ανάλογα με τη διακριτική τη ευχέρεια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ποσοτική ανάλυση αυτή τη τροπολογία λόγω έλλειψη δεδομένων. Τροπολογία 42. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη αναφέρεται σε υποχρέωση σε με τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζεται τακτική και κατάλληλη δικαστική νομική, ε, νομική συνδρομή ή ευεργέτημα της παινίας ε, για ποιον έχει ανάγκη. Επίσης, επίσης, η διάταξη περί νομικής συνδρομής ε, στο κράτος ε, έκδοσης ε, του σχετικού αιτήματο εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και δικαίωμα στην εκπροσώπηση και στο κράτος εκτέλεση και στο κράτος έκδοση απόφαση, συνεργασία για, για να υπάρχουν λιγότερες εσφαλμένες αποφάσεις για την ε, το ευεργέτημα της παινής την λεγόμενη νομική συνδρομή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν στο δυνατόν περισσότερες δυνατότητες για την εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τις δικαστικές αρχές προκειμένου ενδεχομένω ακόμη και να αποσυρθούν ε, εντάλματα βίντεο διάσκεψη περιμένει σε ακροαματική διαδικασία. Αντί ακροαματική διαδικασία. Έτσι αποφεύγονται οι δαπανηρές διαδικασίες και μειώνεται το ανθρώπινο κόστος ε, περίπτωση, δηλαδή να υπάρχει προσωρινή κράτηση ή εσφαλμένη καταδίκη κτλ. Και εδώ μιλάμε για 0,63 1,34 εκατομμύρια ευρώ. Τροπολογία 43 τώρα. Τα κράτη-μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ποιότητα για την παρεχόμενη υπηρεσία, ανεξαρτησία και κατάρτιση των δικηγόρων ε, του βεργηματός της ε, παινίας. Στην τροπολογία 43 δημιουργία ελάχιστων προδιαγραφών ε, σημαίνει ότι θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και τις δεξιότητες οι δικηγόροι που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών ε, με το δικαίωμα σε ελευθερία, στην προσωπική ελευθερία, σε ε, ισότιμη δίκη και στο τεκμήριο της αθωότητας για τον κατηγορούμενο και μείωση του κόστους κατά 13,4 εκατομμύρια για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέτος. Απολογία 44. Δικαίωμα στην έφεση ή προσφυγή κατά της απόφασης αρνηση απόρριψη του αιτήματο της παιγνία ε, και δικαίωμα σε αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα σε περίπτωση που έχει απορριφθεί ή υπονομευθεί ή καθυστερήσει το εν λόγω υπεργέτημα. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα με βάση και το άρθρο 6, τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση για τα κράτη εκείνα στα οποία δεν προβλέπεται μηχανισμός ε, προσβολής απόφασης η οποία απορρίπτει το ετούμενο ευεργέτημα περνίας, ε, οπότε ε, υπάρχει κίνδυνος αυθαιρεσίας ως προς την απόφαση που απορρίπτει. Ε, επίσης θέλουμε να ενισχυθεί ο αριθμός των προσφυγών αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβάρυνση και οικονομική των δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Αλλά δεν είναι το κόστος τόσο σημαντικό, δεδομένου ότι στα περισσότερα των κρατών μελών προβλέπεται το δικαίωμα της προσφυγής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για, τις, ε, για την παρουσίαση και παρακαλώ τους συναδέλφους εφόσον θέλουν να λάβουν το λόγο. Διόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ και τις ερευνήτριες του Μιλίου που ήρθαν για, την, ε, για να μας παρουσιάσουν την ε, μελέτη τους. στο διάλογο για το ευεργέτημα της Περνίας φέτος, στο τριμερή διάλογο μάλλον, είπαμε στο Συμβούλιο, ξεκάθαρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να προωθήσει τώρα και να εξετάσει συνέπειες αλλά και δημοσιονομική διάσταση των προτινωμένων διατάξεων. Θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει έκθεση δική μου, όπου είχα προσπαθήσει να επαναπροσδιορίσω τις προτάσεις περί ευεργετήματος παινίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τις ευθυγραμμίσω με το δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικηγόρο για τον υπόπτωη κατηγορούμενο και τη σχετική οδηγία, ώστε να μην, υπάρχει διαφορά μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των δύο οδηγιών. ή συνέπειε και ο αντίκτυπος νομίζω που καταγράφονται και μέσα από τις τροπολογίες εν γέννη δείχνουν ότι το κόστος που προκύπτει από τις προτάσεις δεν είναι ανυπόφορο, δεν είναι τεράστιο, μάλλον είναι περιορισμένο, όσο δεν αφορά το κέρδος σε προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πρόταση νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία της προτάσεως και έχουμε καταλήξει ένα στάδιο πλέον σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο που έχουμε φτάσει να συνομιλούμε για ε, συμβαστικές προτάσεις κτλ. Ωστόσο, η αξιολόγηση επιπτώσεων είχε την εξή σημασία και συνέπεια ότι για πρώτη φορά ακούσαμε το Συμβούλιο να δηλώνει πως εν γέννη, θα είναι δυνατόν και να καταβάλουμε το κόστος του επιδικομένου στόχου. Αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως είναι περιορισμένο το χρονικό πλαίσιο. Είναι δύσκολο να συλλεγούν για κάθε μία εκ των τροπολογιών επακριβή στοιχεία που θα τις ε, στηρίξουν, όπως είπαν και οι εκπρόσωποι της ε, Ένωσης Μιλίου. Και είδατε κι εσείς ότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Και αυτό είναι και ένας ε, λόγος για τον οποίο έχουμε επικρίνει το Συμβούλιο, γιατί δεν, μπορεί, δεν ήταν σε θέση καν το ίδιο το Συμβούλιο να προσφέρει δεδομένα. Η μόνη παρατήρηση λοιπόν που έχω να κάνω είναι ότι από το ένα κράτος στο άλλο υπάρχουν διαφορές. Κάποια έχουν περισσότερο προχωρήσει στο βαριά τη από ό,τι άλλα. Άλλα λιγότερο. και άρα θα χρειαστούν περισσότερη προσπάθεια για να προχωρήσουν. Αλλά εν γέν θεωρώ χρήσιμη την αξιολόγηση των επιπτώσεων. είναι υπεύθυνο ο τρόπο αυτό εκτέλεση και, των αξιο... και των συνεπειών, τη αξιολόγηση και των συνεπειών. Και όταν έρθει η ώρα, βεβαίω, θα έχουμε στοιχεία, ελπίζω, στη συνομιλία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Ντεϊόγκ. Έτερο. Όχι. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Και κυρίω εδώ πέρα στις συνεδρίαση για την πρωινή μας συνεδρίαση. Στις 3 προβλέπουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Αβραμόπουλο. Επίτροπο μετανάστευση Εσωτερικών και Ιθαγένειας. Καλό μεσημέρι.